Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε καθόλου χρόνο για χάσιμο, πρέπει να ξεκινήσουμε. Ω πρόεδρο τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων, με χαρά καλωσορίζω σε αυτή την ακρόαση τον υποψήφιο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μαργαρίτη Σχοινά. Καλώ ορίσατε, κύριε Σχοινά. Από κοινού με την πρόεδρο τη Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευση, Σαμπίν Φερχάγεν. Η Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι επίση συνδεδεμένη με αυτήν την ακρόαση δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Σύμφωνα με το παράρτημα 7 του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κοινοβουλίο μέσω αυτής της ακρόασης θα αξιολογήσει την γενική επάρκεια, την προσήλωση στο ευρωπαϊκό ιδεώδες και την προσωπική ανεξαρτησία του υποψήφιου επιτρόπου. Επίσης, τη γνώση του χαρτοφυλακίου του και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες. Για την προετοιμασία αυτή της ε, συνάντηση, η διάσκεψη των Προέδρων συνέταξε δύο κοινέ ερωτήσεις, συν έξι ακόμα πρόσθετες ερωτήσεις διαφορετικές για κάθε Επίτροπο. Τρεις από την Επιτροπή ε, Πολιτισμού και τρεις από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ο υποψήφιος Επίτροπος απάντησε στο ερωτηματολόγιο και οι απαντήσει έχουν μοιραστεί. Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν εξέφρασε καμία αντίρρηση στην διεξαγωγή αυτής της ακρόασης. Η συζήτηση θα διαρθρωθεί ως εξής. Ο υποψήφιος Επίτροπος ε, θα κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση για το πολύ 15 λεπτά. Η συνολική ακρόαση θα κρατήσει 3 ώρες το πολύ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ξεπεράσουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά, ερωτήσεις και απαντήσεις για 25 μέλη, 25 βουλευτές, 5 λεπτά για τον κάθε βουλευτή. Ένα λεπτό στην αρχή για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση του υποψηφίου και μετά μια συμπληρωματική ερώτηση από τον ίδιο βουλευτή για ένα λεπτό με απάντηση ενός λεπτού. Συνολικά λοιπόν 5 λεπτά για κάθε ευρωβουλευτή. Ο πρώτος γύρος ερωτήσεων αφορά τους αντιπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Στο δεύτερο γύρο θα έχουμε ερωτήσεις από τους υπόλοιπους βουλευτές συμπεριλαμβανομένων και των μη εγγεγραμμένων. Τέλος, ο υποψήφιος θα έχει στη διάθεσή του πέντε λεπτά για μια τελική τοποθέτηση. Τόσο η κυρία Βερχάγεν όσο και εγώ ίδιος θα είμαστε πολύ αυστηροί σε ό,τι αφορά τον χρόνο αγόρευση. Μη μας αναγκάσετε να σας διακόψουμε παρακαλώ πολύ. Γιατί αλλιώς θα ξεφύγουμε ενώ χρειάζεται να τηρήσουμε τα χρονικά περιθώρια που έχουμε. Διερμηνία υπάρχει σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτή η ακρόαση είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί ο κ. Χινάς ε, είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής που περιλαμβάνει καθοδήγηση και συντονισμό των υποψήφιων επιτρόπων Ήλβα Γιώχανσον εσωτερικών υποθέσεων και Ελένα Ντάλι για την ισότητα που είναι πολύ συναφή θέματα με τα θέματα της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Σχοινά λοιπόν είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, η οποία σύμφωνα με την Συνθήκη της Αβώνας είναι ε, αρμόδια για θέματα ασύλου και μεταναστευτικής πολιτικής, την εσωτερική και την εξωτερική τους διάσταση, το πακέτο ασύλου το πακέτο ασύλου και μετανάστευσης, για παράδειγμα, είναι όπως επίση είμαστε αρμόδιοι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλεια. Οπότε σίγουρα θα προκύψει μια συζήτηση για αυτά ακριβώς τα θέματα και ακόμα και για τον τίτλο του χαρτοφυλακίου. Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής τι ακριβώ σημαίνει. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι υπάρχει ένας ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, αλλά θα πρέπει να δούμε και ποιο είναι το ακριβέ του περιεχόμενο. Τι ακριβώς σημαίνει και ποια είναι, ποιες είναι οι απειλές εναντί των οποίων θα πρέπει να προστατευτεί. Δεν θα πρέπει να κάνουμε κάποια παρανόηση, δεν θα πρέπει να κάνουμε κάποιο λάθος στην ερμηνεία. Γιατί σύμφωνα με τη δική μας άποψη, από την άποψη της Επιτροπής πολιτικών ελευθεριών δεν υπάρχουν απειλέ εναντί του ευρωπαϊκού τρόπου ζωή. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον όλα όσα θα λεχθούν, όπως επίσης ιδιαίτερος για το Σύμφωνο Σύλλου και Μετανάστευσης, το οποίο έχει ανακοινωθεί από την Επιτροπή ότι θα ξεμπλοκαριστεί, όπως ξέρουμε είναι μπλοκαρισμένο στο Συμβούλιο. Θα περάσω τώρα στη, το λόγο στη συμπρόεδρο, την κυρία Φερχάγεν, για τις εισαγωγικές της παρατηρήσεις. Ε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Συμπρόεδρε Λόπεθ Αγγιλάρ για την εισαγωγή σας. Σας ευχαριστώ που παρουσιάσατε πολύ σαφώς πώς ακριβώς θα διεξαχθεί η ακρόασή μας. Από πλευρά τη Επιτροπή για την, τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση, θέλω και εγώ να χαιρετήσω θερμά τον υποψήφιο αντιπρόεδρο, κύριο Σχοινά. Κύριε Σχοινά, είναι πολύ ευρύ το χαρτοφυλακιό σας. Δηλαδή είστε υπεύθυνο για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας και η ευθύνη σας ε, έχει να κάνει και με την μετανάστευση και την ασφάλεια και την απασχόληση και τον πολιτισμό και την, τον αθλητισμό. Σίγουρα δεν θα σας διέφυγε ότι θα υπάρχουν ερωτήσεις για τον τίτλο σας. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης θα έχετε την δυνατότητα να μας παρουσιάζετε την ε, άποψή σας για το πρωτοφόλιό σας. Είναι πολύ θετικό ότι ο συντονισμός ε, της εκπαίδευσης και τον πολιτισμό θα είναι ε, υπό έναν αντιπρόεδρο. Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντική για την Ένωση. Επίσης τίθεται το θέμα πώς ακριβώς θα μεταφραστούν όλα αυτά στην καθημερινή εργασία, ιδιαίτερα στη συνεργασία με την Μαρία Γκαμπριέλ, και για την συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση υπό την αρμοδιότητά της. Εμείς ενδιαφερόμεθα ιδιαίτερα για το πώς θα ε, μπορέσετε να συντονίσετε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και πώς θέλετε να γίνει η εκπαίδευση πιο, πρόσβα, πιο προσβάσιμη και διαμεθοριακή και να συνδυαστεί με την διαβίου κατάρτιση. Και επίσης ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δούμε με τι μέσα θα χρησιμοποιήσετε για να μπορέσουν να ενταχθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Ορισμένα βασικά σημεία είδαμε στην ε, γραπτή σας απάντηση. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις απαντήσεις που δώσατε. Και με πολύ προσοχή θα ακούσω κατά τις επόμενες τρεις ώρες ε, την άποψή σας για τους διάφορους τομείς πολιτικής για τους οποίους είστε αρμόδιος και είμαι σίγουρη ότι η ακρόαση αυτή θα δώσει απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Οπότε προσβλέπω σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας κύριε και να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Φερχάιεν και κύριε Πρόεδρε λόπεθα Αγγιλάρα. Αξιότιμα μέλη. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη στιγμή για μένα αυτή και έχει μεγάλη συναισθηματική φόρτιση τα τελευταία 30 χρόνια σε αμέτρητες ε, στιγμές είχα δυνατότητα να συμμετάσχω σε μια σειρά από επιτροπές και άλλα όργανα του σώματός σας. Πρώτα ως νέος υπάλληλο, μετά ως τέλεχος και αργότερα ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά άλλη διάσταση έχει τώρα η σημερινή συμμετοχή μου. Είμαι εδώ τώρα, ενώπιόν σας, ως υποψήφιος αντιπρόεδρος, ζητώντας την εμπιστοσύνη σας, ούτως ώστε να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα εργασιών για τα επόμενα πέντε χρόνια μαζί σας. Συναισθάνομαι πραγματικά το βάρος των ευθυνών μου. Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση μας υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε μια κοινωνία στην οποία ο πλουραλισμός, η έλλειψη διακρίσεων, η αποδοχή των άλλων, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι τα κυρίαρχα στοιχεία. Με αυτή τη διατύπωση η συνθήκη για μένα καθορίζει σαφέστατα την αποστολή μου ως Αντιπροέδρου. Το χαρτοφυλάκιό μου, οι αρμοδιότητές μου έχουν να κάνουν από την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την απασχόληση, την ασφάλεια, την μετανάστευση, μέχρι την υγεία και την ισότητα αλλά το κοινό νήμα όλων αυτών των ε, τομέων πολιτικής είναι οι συμπολίτες μας. Πρέπει να υπερασπιστούμε την απλή αλλά ουσιώδη προϋπόθεση ότι όλοι μετράνε, ότι δεν θα πρέπει να γνωριθεί κανείς, ότι όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ίδια δικαιώματα, την ίδια ασφάλεια, τις ίδιες ευκαιρίες. Αυτή είναι η βασική αρχή η αφετηρία μου, εάν με επιβεβαιώσετε ως Αντιπρόεδρο. Θεωρώ ότι ο συντονιστικό μου ρόλος θα έχει μια σημαντική προστιθέμενη αξία σε τρεις κυρίους τομείς, όπου θα επικεντρώσω τη σύντομη εισαγωγική μου ομιλία. Πρώτα απ' όλα, να κάνουμε τις κοινωνίες μας δικαιότερες, που να συμπεριλαμβάνουν περισσότερους συμπολίτε μας. Δεύτερον, να έχουμε αποτελέσματα για ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, και τρίτον να ολοκληρώσουμε την ε, Ένωση Ασφάλειας για να αντιμετωπίσουμε τους παραδοσιακούς αλλά και τους, ε, τις παραδοσιακές αλλά και τις απειλές της σύγχρονης εποχής. Σε όλους αυτούς τους τομείς τα μέτρα που πρέπει να λεφθούν πρέπει να ε, ξεπεράσουν τα οργανωτικά στεγανά. Η δουλειά μου θα είναι να συνδυάσουμε την εμπειρογνωμοσύνη από όλους τους τομείς πολιτικής και να εστιάσουμε στους συμπολίτε μας και σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου τη συζήτηση που προκλήθηκε από τον τίτλο που δόθηκε σε αυτή την εργασία. Έχω κάθε σεβασμό για όλες τις θέσεις που εκφράστηκαν και όλα τα επιχειρήματα που εκφράστηκαν σε αυτή τη συζήτηση. Σύμφωνα με τον Σέξπιερ, ένα ρόδο, όπως και να το ονομάσεις, θα έχει την ίδια γλυκιά μυρουδιά. Αλλά τα ονόματα είναι σημαντικά. Γιατί δίνουν έννοια στα πράγματα. Δίνουν και σε εμά έννοια. Και κάτι σημαίνει το να είσαι Ευρωπαίος. Στον πυρήνα της, η έννοια του Ευρωπαίου σημαίνει προστασία των πιο ευαλώτων ε, στις κοινωνίες μας. Σημαίνει υγεία και συστήματα πρόνοιας προσβάσιμα σε όλους σημαίνει να έχουμε όλοι τις ίδιες ευκαιρίες. Σημαίνει προώθηση του πολιτισμού και του αθλητισμού που είναι βασικά στοιχεία του συστήματός μας. Σημαίνει να δώσουμε σε όλους τους συμπολίτε τη γνώση, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζήσουν και να εργάζονται με αξιοπρέπεια. Σημαίνει να αισθανόμεθα ασφαλείς στα σπίτια μας, στους δρόμους μας και σε όλους τους τόπους όπου συναντιόμαστε, συζητάμε, και έχουμε κοινέ εμπειρίε ζωή. Ευρωπαίο σημαίνει επίση να είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο. Να ανοίγουμε την καρδιά μα και το σπίτι μα στου λιγότερο τυχερού από εμά. Σημαίνει να προωθούμε αυτά τα ίδια δικαιώματα, τι ίδιε αξίε και αρχέ παντού στον πλανήτη. Ευρωπαίο σημαίνει ελευθερία, ειρήνη, ισότητα, δημοκρατία και σεβασμός για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και κάτι πολύ προσωπικό. Για μένα Ευρωπαίος σημαίνει ότι έχω ζήσει στην Ευρώπη, ότι έχω μεγαλώσει την οικογένειά μου στην Ευρώπη και ότι έχω αφιερώσει 30 χρόνια της ζωής μου στην ε, υπηρεσία της Ευρώπης ως δημοσίου λειτουργού. Είμαι πρώτα και κύρια Ευρωπαίος και είμαι περήφανος που είμαι Ευρωπαίος ακόμη πιο περήφανος γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα να υπηρετήσω αυτήν την Ένωση. Αξιότιμα μέλη. Οι επιτροπές που εκπροσωπούνται εδώ σήμερα είναι ηγέτες στην προσπάθεια οι κοινωνίες μας να συμπεριλάβουν περισσότερους συμπολίτε και να είναι πιο ανθεκτικές. Και πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον που να βασίζεται στην πρόσβαση για όλους και στις ευκαιρίες για όλους. Να ξεκινήσω με το πρώτο κεφάλαιο των παρατηρήσεών μου. Πώς θα κάνουμε τις κοινωνίες μας δικαιότερες, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους συμπολίτε. Είναι γνωστό ότι οι κοινωνίες μας προστατεύουν τους πιο ευάλωτους μεταξύ ημών. Και αυτό θέλω να ισχύει για όλους. Εάν ε, με βεβαιώσετε, θα χρησιμοποιήσω τις αρμοδιότητές μου σε πολλούς τομείς, ούτως ώστε να έχουμε μια συνολική αντίληψη για ακριβώς τη συμπερίληψη και την ένταξη. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ήταν ορόσημο. Αλλά πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα δικαιώματα και οι αρχές θα ε, γίνουν καθημερινή πραγματικότητα. Ένα από τα κύρια καθήκοντά μου θα είναι να διασφαλίσω ότι το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ θα βοηθήσει την ένταξη, θα στηρίξει αυτού που έχουν ε, τι μεγαλύτερε ανάγκε και θα βοηθήσει να υπάρξει περισσότερη κινητικότητα των εργαζομένων παντού στην Ένωση. Πρέπει η νεολαία μα να έχει τις σωστές δεξιότητες για να προκόψει στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. Θα εργαστούμε ούτω ώστε ο Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευση να γίνει πραγματικότητα. Θα δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη για να μεταρρυθμίσουν και να εξυγχρονίσουν τα συστήματα εκπαίδευση και κατάρτιση. Εμένοντα στην ψηφιακή κατάρτιση, θα διασφαλίσω ότι θα αξιοποιήσουμε το Erasmus In, το Discovery U και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη, ούτω ώστε να δώσουμε περισσότερε δυνατότητε στου νέου μα και να τους δώσουμε νέες δυνατότητες κινητικότητας. Να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αφήνουμε πίσω κανένα παιδί. Γι' αυτό θα εισαγάγουμε την εγγύηση, την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, ώστε τα παιδιά που κινδυνεύουν από αποκλεισμό και φτώχεια να έχουν πρόσφαση στα βασικά δικαιώματα όπως είναι η υγεία και η εκπαίδευση. Αυτό είναι κάτι που το ξεκινήσατε εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Και αυτή την δέσμευση θα την τηρήσουμε. Θα εργαστώ με την Επίτροπο για την Υγεία, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά συστήματα υγεία ε, δεν θα ξεχνούν κανένα και θα συνεργαστώ με την Επίτροπο για την Ισότητα, ούτω ώστε να υπάρχει ισότητα σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των φύλων και θα πιέσουμε για να προχωρήσει η νομοθεσία κατά των διακρίσεων και η Ευρωπαϊκή Στρατηγία το φύλλο, που θα προωθήσουν την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Αυτή η νέα προώθηση τη συμπερίληψη σε όλου του τομεί θα πρέπει να, να συμπεριλάβει και μια νέα όθηση για την ένταξη των υπηκών τρίτων χωρών θα εργαστώ με βάση το σχέδιο δράση του 2016 για την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών, ούτω ώστε να υπάρξουν συμπληρωματικοί πόροι. Χαίρομαι που η μακροπρόθεσμη ένταξη των μεταναστών και προσφύγων θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Αυτό θα μα επιτρέψει να έχουμε περισσότερα μέσα στη διάθεσή μα και περισσότερου πόρου για να στηρίξουμε αυτέ τι πρωτοβουλίε. Και να μην ξεχνάμε ένα από του θησαυρού τη Ευρώπη είναι η πολιτιστική μα κληρονομιά. Πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτήν και να την προωθούμε εντό και εκτό τη ένωση. Αλλά και ο αθλητισμός μπορεί να έχει θετική επίπτωση στην κοινωνία για την υγεία, την ένταξη και την ισότητα των φίλων. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τι κοινωνίε μα και τι οικονομίε μα ε, να πάνε καλά, πρέπει να στηρίξουμε όλου του συμπολίτε μα, όλου που είναι τμήμα ακριβώ των κοινωνιών. Η συμπερίληψη όλων είναι και δικαιώμα αλλά και υποχρέωση για όλους μας. Τώρα να στραφώ στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας μου, δηλαδή πώς θα έχουμε ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Αυτό είναι δυσχερές έργο, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να το επιτύχουμε εάν αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε και μαθαίνοντας από το παρελθόν. Αυτό το νέο σύμφωνο πρέπει να καλύπτει πολλούς τομείς και να συνδυάζει τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές η μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ευρωπαϊκού ασύλου. Εδώ το πρώτο που θα κάνουμε μαζί με ε, την Επίτροπο για τις Ιστορικές Υποθέσεις είναι να ξεκινήσουμε διάλογο μαζί σας και τα κράτη-μέλη. Πρέπει να βρούμε ακριβώς που υπάρχει περιθώριο για συμβασμούς. Θα ακούσουμε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Θα σας ε, παρουσιάσουμε σύντομα εναλλακτικέ λύσεις, τις οποίες θέλουμε να συζητήσουμε, για να βρούμε συνένεση. Αλλά μόνο τότε θα κάνουμε επίσημες προτάσεις. Μετά από τα προηγούμενα λοιπόν. Δεν θα αμελήσουμε καθόλου την τεράστια εργασία που έχει ήδη επιτελεστεί τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και τους συμβασμού που έχουν ήδη εξευρεθεί σε πολλά τμήματα του πακέτου για τη μεταρρύθμιση του ασύλου. Όλα αυτά ξέρω πολύ καλά. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό χάρη σε εσά, εδώ στο Κοινοβούλιο. Όλα αυτά θα τα διατηρήσουμε. Οι εσωτερικές μας μεταρρυθμίσει, ωστόσο, είναι μόνο τμήμα μιας πολύ ευρύτερης εικόνας. Ως προσωρινή λύση, μέχρι να υπάρξει ένα νέο και πραγματικά κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη μέσω προσωρινών διευθετήσεων για τον, την αποβίβαση. Για μένα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε και σωστό διάλογο με τις πολλές μη κυβερνικέ οργανώσεις που κάνουν αξιόλογη δουλειά για την έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο πρέπει και αυτές να είναι τμήμα της λύσης. Όλες σήμερα που είναι τραγική επέτειος ε, της ε, τραγωδίας της ε, Λαμπεντούζα, αυτό είναι πολύ πιο αναγκαίο από ό,τι προηγούμενα. Όλες οι προτάσεις και πρωτοβουλίες του νέου συμφώνου θα γίνουν με τον παράλληλο στόχο να αρθούν οι εσωτερικοί έλεγχοι στα σύνορα, ούτως ώστε να επανέλθουμε σε μια πλήρη λειτουργική περιοχή Σέγγεν ένα αξιόπιστο σύστημα ασύλου επίσης πρέπει να προστατεύσει από την κατάχρηση του συστήματος. Θα είμαι επικεφαλής μιας νέας προσπάθεια να υπάρξουν επιστροφές για αυτούς που δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν. Πρώτα απ' όλα συμπληρώνοντα τη μεταρρύθμιση των εσωτερικών μας κανόνων για τις επιστροφές και δεύτερον συνάπτοντας συμφωνίες επανεισδοχής και διαδικασίες με τις χώρες προτεραιότητας, διέλευση και προέλευση. Πρέπει επιτέλους τώρα να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα για να στηρίξουμε τι προτεραιότητες μα στα θέματα αυτά. Τέλο, πρέπει να κάνουμε περισσότερα με βάση τα πιλωτικά προγράμματα για την νόμιμη μετανάστευση. Τα πιλωτικά ήδη έχουν ξεκινήσει. Θέλουμε σύγχρονε και στοχευμένε ε, προτάσει για την νόμιμη μετανάστευση που να ανταποκρίνονται στι ανάγκε τη οικονομία μα, τη αγορά εργασία μα και των δημογραφικών προκλήσεων. Και θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι με βάση το μοντέλο των ε, μηχανισμών επίγουσας ανάγκης ε, με το Νίγηρα και τη Ρουάντα τώρα. Τέλος. Οι ευθύνες μου τώρα για την ε, Ένωση Ασφαλείας. Οι αξίες της Ευρώπης δεν πρέπει μόνο να αναφέρονται, αλλά να διασφαλίζονται έναντι των απειλών του. Η Ένωσή μας είναι ε, πρωτοπόρα στην προστασία των δεδομένων και του ιδιωτικού βίου και είμαι, έχω κάθε συνέστηση ότι αυτά που κάνουμε για την ασφάλεια πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο σεβασμό των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να είναι τμήμα από την αρχή αυτών των πολιτικών. Αυτό θα είναι οδηγό μου και στην εργασία μου για να εφαρμόσουμε τι προτάσει για την διαλειτουργικότητα που θα είναι πολύ σημαντικέ γιατί ξεκινάμε για να εφαρμόσουμε νέα συστήματα πληροφοριών. Επίσης, θα ασχοληθώ αδιάκοπα με την εφαρμογή όσων αποφασίζουμε. Θα προωθήσω μια συντονισμένη προσέγγιση για να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους στο ίντερνετ μέσω της έγκρισης της πρότασης για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο ίντερνετ και συμβάλλοντας ε, στην πράξη για τις ε, ψηφιακές υπηρεσίες και εργαζόμενοι και μέσω του ενωσιακού φόρουμ για το ίντερνετ. Θα αξιοποιήσω όλες τις δυνατότητες που έχω για να έχουμε καλύτερη ανταπόκριση στις υβριδικές απειλές που απειλούν τα συστήματά μας, ακόμη και την δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, υπήρξα μέλος ε, του Κοινοβουλίου και ξέρω πολύ καλά ότι η καρδιά της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας είναι εδώ. Εδώ ε, εγκρίνονται οι νόμοι μας. Εδώ διαμορφώνεται το μέλλον μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξελέγει με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό αποδεικνύει την ενεργό δέσμευση των συμπολιτών μας που συμμετέχουν και δεν δίνουν μορφή στη δημοκρατία μας. Δεν μπορούμε να τους απογοητεύσουμε. Για μένα αυτό σημαίνει ότι έχω την πλήρη ευθύνη έναντί σας ότι θα υπάρξει μεγάλη διαφάνεια όσον αφορά την εργασία μου και το άτομό μου. Κλείνω λέγοντας ότι δεσμεύομαι να εφαρμόσω τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και διαφάνειας με σεβασμό στη συνθήκη και τον κώδικα συμπεριφοράς των επιτρόπων, δεσμεύομαι να εργαστώ συλλογικά με τους συναδέλφους μου και να εργαστώ ακούραστα μαζί σας για μια ένωση ασφαλέστερη για τους πολίτες μας, πιο ισότιμη, χωρίς αποκλεισμούς. Πάνω απ' όλα δεσμεύομαι με όλες τις δυνάμεις μου να θέσω ως απόλυτη προτεραιότητα τους ανθρώπους. Πέρα και πάνω από κομματικές γραμμές και εθνικά σύνορα, η δική μας Ένωση πρέπει να είναι μια Ένωση ανθρώπων. Μια Ένωση στην οποία κανένας δεν θα βρίσκεται στο περιθώριο. Μια Ένωση πολιτών που ζουν σε συνεκτικές και ανεκτικές κοινωνίες. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Σκινά. Περνάμε στο πρώτο μέρο, στο πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Ο πρώτο γύρο των ερωτήσεων, 7 θα είναι, οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Ξεκινάμε με την Ρομπέρτα Μετσόλα για το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Ευχαριστώ υποψήφια την Πρόεδρε για την διεξοδική σας παρουσίαση. Το ΕΛΚ καλωσορίζει το γεγονός ότι το χαρτοφυλάκιό σας θα αγγίζει πολλά, θε, πολλές διαστάσεις αλληλένδετες του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Διότι όπως είπατε το χαρτοφυλάκιό σας αφορά τελικά τους ανθρώπους. Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής εδράζεται στις συνθήκες. Στις συνθήκες. Ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, η πολυφωνία, η μη διακριτική μεταχείριση, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη. Είμαστε υπερήφανοι για τι αξίε αυτέ, και υπερήφανοι και για το παράδειγμα που δίνουν όχι μόνο στους Ευρωπαίου, αλλά σε όλο τον κόσμο. Το χαρτοφυλάκιό σα απαιτεί να αναλάβει κανεί ε, ηγετικό ρόλο και αυτό περιμένουμε από εσά. Πώ σκοπεύετε να διασφαλίσετε ότι η ισότητα και η ποικιλομορφία που είναι τόσο πολύ μέρο του τρόπου ζωή μα, θα ενισχυθούν. Πώ θα βεβαιωθείτε ότι η συμπερίληψη και η ένταξη θα παραμένουν ακρογωνίως λίθος της δουλειάς σας και πώς θα συντονίσετε τα του νέου συμφώνου μετανάστευσης προκειμένου να παραμένουν ε, συνεκτικές οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς και η εσωτερική και εξωτερική διάσταση. Ευχαριστούμε κυρία Μετζόλα. Κύριε υποψήφια, Επίτροπε, Αντιπρόεδρε, δύο λεπτά για την απάντησή σας. Για τις αξίες και το πώς αυτές οι αρμοδιότητες που άπτονται πολλών τομέων ταυτόχρονα και πώς αυτό μπορεί να εμπλουτίσει τη δουλειά μας για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε, το πώς μπορεί να συνδυάσουμε τις νέες ανάγκες που θα παρουσιαστούν στις κοινωνίες μας, τις δεξιότητες, τις θέσεις εργασίας, τη μετανάστευση. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι προφανή. Δεν χρειάζεται να πω πολλά λόγια. Ε, έχουμε πετύχει αρκετά εργαζόμενοι σε αυτήν την κατεύθυνση προς τώρα. Τώρα όμως πρέπει να ε, κοιτάξουμε τους καρπούς όλων αυτών των παράλληλων ε, δρόμων κατευθύνσεων εργασίας για να παράγουμε νέες αξίες και νέα αποτελέσματα. Χαίρομαι και πραγματικά ενθουσιάζομαι με αυτές τις νέες μου αρμοδιότητες, διότι έχει να κάνει με τη συνεργασία με τους άλλους επιτρόπους και με εσάς εδώ, με όλους από τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά το σύμφωνο, ένα από τα μαθήματα που μπορούμε να αντλήσουμε στο χώρο αυτό μαζί με τη συνάδελφό μου την Ήλβα, χρειαζόμαστε σαφώς μια νέα αρχή. Αυτό είναι το κυριότερο. Πρέπει να ξαναδούμε τι δεν πήγε καλά στο παρελθόν και δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Χωρίς να ξεχάσουμε τις πέντε ε, βασικές μας, τα, τα πέντε βασικά σημεία που έχει γίνει ήδη μεγάλη πρόοδος, σοβαρή πρόοδος. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο σημείο που θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο συμφωνό, δηλαδή στον, στην αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου και των σχετικών κανόνων, αλλά θα πρέπει να συνδέσουμε με αυτή την προσπάθεια οτιδήποτε χρειάζεται για να ε, ξεπεράσουμε την ε, δυσκολία στην οποία έχουμε βρεθεί, για να ε, είναι σαφής και σφαιρική εικόνα για όσους έχουν μια μερική εικόνα του τι πρέπει να γίνει ως τώρα. Ε, και τώρα δεύτερη ερώτηση για την κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση συγκεκριμένα, ενώ οι αφήξει έχουν μειωθεί, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που χάνουν στις ζωές τους τις ακτές μας. Τα δίκτυα των εμπόρων ανθρώπων ακόμα λειτουργούν και οι επιστροφές δεν έχουν φτάσει στα ύψη που θα θέλαμε και στο ρυθμό που θα θέλαμε. Δεν υπάρχει ένα σύστημα κατανομής των ευθυνών, οι χώρες προέλευσης ακόμη χρειάζονται περισσότερο περισσότερε ευρωπαϊκέ επενδύσει για να στηρίξουν τα συστήματά του και συμφωνίε επανεισδοχή δεν έχουν προχωρήσει. Σαφώ χρειάζονται περισσότερα. Τι μπορείτε όμω εσεί να κάνετε με διαφορετικό τρόπο την ερχόμενη πενταετία. Πράγματα που δεν έχουν δοκιμαστεί ή πράγματα που έχουν ε, μπλοκαριστεί σε άλλο επίπεδο. Τι μπορείτε να κάνετε από την πλευρά των αρμοδιοτήτων σα και ω προ την νόμιμη μετανάστευση. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν πρέπει όμω να γίνει μια σοβαρή αξιολόγηση ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι δεξιότητε λείπουν από τα κράτη-μέλη και να τι συνδυάσουμε με όσου παρανόμω αφικνούνται στα κράτη-μέλη. Ε, κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε, δύο λεπτά. Ένα λεπτό. Να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα στην πρώτη σας ερώτηση. Νομίζω θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση στην αναθεώρηση του κανονισμού του Δοβλίνου ε, και τι σχετικέ διαδικασίες. Θα πρέπει η κατάσταση να απεμπλακεί ώστε να συνδυάσουμε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία και να έχουμε μια συνολική εικόνα. Ε, επιστροφές, νέε ναι, συμφωνίε επανεισδοχή, Σέγγεν, σύνορα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο να δει ότι δεν υπάρχει μία συνιστόσα ή ένα θέμα που μπορεί να είναι η μαγική λύση σε όλα αυτά. Πρέπει όλα μαζί ταυτόχρονα να τα δούμε ε, και εσωτερικός και εξωτερικός. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να δούμε τι χρειάζεται και μετά να καλέσουμε κόσμο να έρθει. Και για την νόμιμη μετανάστευση θα πρέπει να βασιστούμε στην επιτυχία των πιλωτικών προγραμμάτων, να ξαναδούμε την οδηγία για τη γαλάζια κάρτα, την πρόταση για τη γαλάζια κάρτα που έχουμε επιτάπητος και με όσο περισσότερο ευθύ τρόπο μπορούμε να δούμε αν υπάρξει αντιστοίχηση των δημογραφικών μας αναγκών και των δεξιότητων που λείπουν με νόμιμες διόδους, νόμιμες ε, οδούς. Ευχαριστούμε. Και τώρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες η κυρία Σίπελ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Σκηνά. Δυστυχώς ο τίτλος του χαρτοφυλακίου σας ε, έχει γίνει παιχνίδι στα χέρια των ε, ακροδεξιών και σαν να φαίνεται ότι δημιουργούμε το χειρό Ευρώπη. Η μετανάστευση είναι μια πρόκληση, αλλά οι μετανάστες δεν είναι απειλή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από διώξηση, αναζητούν εργασία. Αυτό είναι τμήμα και της δικής μας ιστορίας. Στην δική σας επιστολή λέτε ότι πρέπει να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή μας κουλτούρα. Από ποιον θα πρέπει να την προστατεύσουμε και μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι το χαρτοφυλάκιό σας δεν θα προσπαθήσει να ομογενοποιήσει τη, θε, τη θεώρησή μας, αλλά ότι θα είναι ε, μια αρχή για να συμπεριλάβουμε όλους και να μην αφήσουμε κανέναν εκτός. Minutes for answer, Vice President Δύο, δύο ε, λεπτά για την απάντηση. Ο κ. Σχοινά. Ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί μου επιτρέπει να διευκρινίσω κάτι. Προσπάθησα να κάνω βέβαια και στις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις. Εγώ ποτέ, ποτέ δεν συμμερίστηκα την άποψη ότι ο τίτλος του χαρτοφυλακίου μου μπορεί να οδηγήσει στο να πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε σε αντίθεση, σε σύγκρουση με κάποια άλλη κουλτούρα. Όχι, που δεν είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας φάρος, φωτεινός φάρος σε ένα κόσμο που σκοτεινιάζει. Έχουμε ποικιλομορφία, είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας, είμαστε ιδιαίτεροι, μας θαυμάζουν και μας ζηλεύουν. Και είναι και προς δικός μας όφελος να χρησιμοποιήσουμε με θετικό τρόπο αυτά τα χαρακτηριστικά μας, να κάνουμε μια πιο ανθεκτική κοινωνία χωρίς να φοβόμαστε και να αυτομαστιγωνόμαστε, να μην χρειάζεται να ζητάμε συγγνώμη για τις αρχές μας και τα ιδεώδη μας. Και κάποιοι λαϊκιστές μπορεί να προσπαθούν ε, ε, να εργαλειοποιήσουν τις αρχές μας, αλλά οι αρχές μας είναι πάρα πολύ ανθεκτικές και δεν απειλούνται από τους λαϊκιστές. Οι λαϊκιστές θα πρέπει να αισθάνονται απειλούμενοι από τις αρχές μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια εχθρικότητα. Οι μεταναστευτικές μας πολιτικές δεν κάνουν εξαιρέσεις, δεν κάνουν αποκλεισμού και βασίζονται στην υπόθεση εργασία ότι θα εξακολουθήσουμε να είμαστε μια περιοχή η οποία θα δέχεται μετανάστευση. Αυτή αυτό είναι ο χαρακτήρας μας, αυτή είναι η φύση μας. Η Ευρώπη πάντοτε θα είναι μια περιοχή που θα δέχεται μετανάστες και ε, θα δίνει άσυλο. Αυτοί όμω οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψουν και αυτό θα γίνει. Με το δικό μας ευρωπαϊκό τρόπο πάλι, σύμφωνα με τις δικές μας αρχέ, με ένα ανθρώπινο τρόπο, με αξιοπρέπεια και με δικά μας χρήματα. Με μετριοπάθεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό θα πρέπει να μας κάνει να αισθανόμαστε ένοχοι ή να ζητούμε συγνώμη. Θέλω να τονίσω τη θετική πλευρά όλων αυτών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζίπελ. Για ένα λεπτό συμπληρωματική ερώτηση. Δυστυχώς δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου έναντι ποιον προστατεύουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή μας και πώς θέλετε να προωθήσετε τις αρχές μας και την κουλτούρα του κράτους δικαίου. Δεσμεύεστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστεί υπέρ μια Ευρώπη που θα τίνει χείρα σε αυτού που βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη αλλά και σε αυτού που θα έρθουν. Τι ακριβώ το καινούριο θα έχει το καινούριο σύμφωνο μετανάστευση, σε τι θα διαφέρει από την υπάρχουσα νομοθεσία και τι προτεραιότητε θα έχει θα διαφέρει από την ε, πρόταση του Κοινοβουλίου για μια ολιστική σφαιρική αντιμετώπιση τη μετανάστευσης. Σε ό,τι δεν αφορά τον τίτλο, δεν είπα ότι εσείς συμμερίζεστε την αρνητική ερμηνεία του τίτλου. Παρόλα αυτά, αυτή η ερμηνεία γίνεται, υπάρχει. Και στις γραπτές ερωτήσεις σας ρωτήσαμε αν είστε διατεθειμένο να αλλάξετε τον τίτλο, δεν μα απαντήσατε. Οπότε δεσμεύεστε να αλλάξετε τον τίτλο του χαρτοφυλακίου σας. Ένα λεπτό για τον κύριο Σχοινά. Να ξεκινήσω με το ε, έναντι ποιου προστατεύουμε τον τρόπο ζωής μας. Έναντι αυτών που δεν μας επιτρέπουν να γιορτάζουμε τη 14η Ιουλίου στην Ίκαια. Έναντι αυτών που δεν μας επιτρέπουν ε, να εργαζόμαστε στις Ράμπλα στη Βαρκελόνη. Έναντι αυτών που αντί να βοηθούν τους μετανάστες, τους χώνουν σε ένα στρατόπεδο, σε ένα καταβλισμό έναντι αυτών που δεν θέλουν να δίνουμε φαΐ στους ετούντες άσυλο, που δεν θέλουν να επιτρέψουμε στα παιδιά τους να πηγαίνουν στο σχολείο. Έναντι αυτών των στοιχείων θέλουμε να προστατευτούμε. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όμως αυτές τις προκλήσεις με θετικό τρόπο, χωρίς αποκλεισμού. Και επαναλαμβάνω ότι επουδενή η δική μου θεώρηση αυτού του χαρτοφυλακίου που δημιουργείται για πρώτη φορά τώρα ασφαλώς, επουδενή η θεώρησή μου δεν θα είναι αρνητική. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι λαϊκιστές θέλουν να το εκμεταλλευτούν, αλλά δεν θα πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι τους. Δεν θα είναι αυτός ο ρόλος μου. Σε ό,τι αφορά το σύμφωνο, νομίζω ότι ήμουν πολύ συγκεκριμένος στην απάντησή μου στην κυρία Μετσόλα. Αν θέλετε θα μου δώσετε περισσότερες ευκαιρίες να εξηγηστώ. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στην ομάδα Renew. Η κυρία Ιντβελτ, ένα λεπτό για την ερώτησή σας. Ευχαριστώ, υποψήφια Επίτροπε. Πρέπει να πω ότι δεν έχω καμία αμφιβολία για την προσωπική σας αφοσίωση και ότι είστε ταγμένος στις αξίες που εξηγήσατε. Όμως, πραγματικά, ε, κάνατε και μια προσπάθεια να υπερασπιστείτε τον τίτλο σας που είναι ματή. Δεν μπορεί κανείς να τον προασπιστεί. Τι θα πει προστατεύουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας. Ε, είστε πολύ ε, έμπειρος ε, στα επικοινωνιακά και νομίζω ότι κατανοήσατε ευθύ αμέσω. Ο τίτλος αυτός συνδυαζόμενος με το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης έχει τοξικό χαρακτήρα. Ε, είναι μια νίκη της ακροδεξιάς αυτή η έκφραση. Ξέρετε ότι καμία ερμηνεία και καμία εξήγηση δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Είναι σαφές ότι η κυρία Φοντελάιν έχει εμείνει ως τώρα. Και βεβαίως όποια προσπάθεια έγινε να ενωθούν εδώ οι απόψει τελικά δεν το πετυχαίνει γιατί δείχνει ότι θα αποκλειστεί κόσμο και προκαλεί διχασμού. Βλέπω ότι πολλοί χαιρόνται οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ. Το ΕΛΚ ε, είναι σε θέση να ελέγχει τι αντιδράσει του, αλλά με μισή καρδιά και χαιρέται η ακροδεξιά. Δεν ήταν λάθο η επιλογή του τίτλου αυτού, ή μήπω και χειρότερα, δεν ήταν μια κακή πολιτική κρίση τελικά. Κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε, δύο λεπτά. Κυρία Ιντφελτ, ξεκινώ από την ε, αρχή ότι σέβομαι όλα τα επιχειρήματα και όλες τις τοποθετήσεις που εκφράζονται στη συζήτηση περί του τίτλου μου. Καμία αντίρρηση από αυτού ε, και δεν έχω κάτι να πω εναντίον της οποιασδήποτε άποψη εκφράζεται. Ωστόσο, και όταν διάβασα και το άρθρο που έγραψε σε μια εφημερίδα ευρωπαϊκή πολύ γνωστή πριν από λίγες εβδομάδες η ε, πρόεδρος, η πρόεδρος ε, και είπε πώς βλέπει τη σχέση των χαρτοφυλακίων με τα άρθρα της Στο άρθρο αυτό υπάρχει μια τελική παράγραφος, μια τελευταία παράγραφος που λέει ότι μέρος του ευρωπαϊκού μας τρόπου ζωής είναι ακριβώς ότι στην Ευρώπη πάντοτε συζητούμε και μετά συμφωνούμε βρίσκουμε συμφωνίες. Εφόσον λοιπόν ε, με προκαλείτε να τοποθετηθώ εγώ απέναντι σε αυτό το γεγονός, πρέπει να πω ότι έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ε, κυρία Φοντερ για το επιχείρημα αυτό. Ε, είναι έμπειρη στο κοινοβουλευτικό βίο, όσο και εσείς, και Νομίζω μεταξύ του σεβασμού όλων των επιχειρημάτων που εκφράζονται και τη δική της την επιθυμία και προθυμία να αφουγκραστεί, να ακούσει και να, βρε, να, να εξεύρει συμφωνίες, νομίζω ότι ουσιαστικό μας οδηγεί στο ότι ο χρόνος θα δώσει την απάντηση που τώρα εσείς μου ζητάτε. Okay, over to... Ωραία. Και πάλι εσείς κυρία Ιντφελτ για την επερώτησή σας. ενδιαφέρον. Έχουμε δύο λεπτά νομίζω. Έτσι κι αλλιώς. Διότι η ερώτηση, ε, πραγματικά και σοβαρά τώρα, δεν αφορά εσάς προσωπικά, ε, αλλά και όλη την Επιτροπή και την κυρία Φαντερ Τι ακριβώς θέλει να πετύχει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, διότι ήταν πολύ μικρή η πλειοψηφία με την οποία πέρασε η πρόταση τον Ιούλιο. Και εδώ καλό θα ήταν να έχουμε μια στενή σχέση με το Κοινοβούλιο και όχι ένα μεγάλο σοου για το πόσο φοβερός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Ε, και μπορεί να είναι καλύτερο να ε, έχουμε μια ε, προσέγγιση του κέντρου παρά κάτι διαφορετικό. Πιστεύει η ομάδα μου ότι ο τίτλος πρέπει να αλλάξει, πρέπει να, να φύγει και πραγματικά ας αφήσουμε αυτή την προσπάθεια να τον υπερασπιστούμε και τα επόμενα πέντε χρόνια κοιτάξουμε να φτιάξουμε μια Ευρώπη ε, που θα συμμετέχουν όλοι, που θα είναι για όλους. Διότι η Ευρώπη θέλουμε να είναι παγκοσμίω πρωταθλήτρια της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της αλληλεγγύης. Εσείς πρέπει να κάνετε την επιλογή κύριε Σχοινά θα ε, πάρετε και σε θέση ώστε ο τίτλος αυτός να αλλάξει και να φύγει. Είτε κερδίζετε, είτε... Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να ξαναρχίσουμε το χρονόμετρο. Διότι έπεσαν χειροκροτήματα μόλις ξεκινήσαμε το λεπτό. Ένα λεπτό από τώρα, κύριε Σκηνά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν η κυρία Φαντρελάιεν υπέβαλε τι προτάσει τη για τι πολιτικέ τη γραμμέ τον Ιούλιο στο Κοινοβούλιο. Πρότεινε έξι βασικέ κατευθύνσει για τη δουλειά που πρότεινε να γίνει γραπτό και στην ομιλία τη. Μία από αυτέ ήταν η προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωή. Το περιεχόμενο εξηγήθηκε νομίζω με σαφήνεια. Και πήρε την ψήφο εμπιστοσύνη ε, του σώματος αυτού. Είναι υποψήφια πρόεδρος, διότι της αποδώσατε την εμπιστοσύνη σας βάσει αυτών των έξι κατευθυντηρίων γραμμών, οι οποίες, των οποίων λάβατε γνώση και τις εγκρίνατε. Καταλαβαίνω ότι έκτοτε έχουν συμβεί πολλά βέβαια και καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε εδώ κάπως να παντρέψετε τις αρνητικές εντυπώσεις, προδικάζοντας το τι δουλειά θα κάνω εγώ, ενώ έχω ήδη αφιερώσει χρόνο στο να σας εξηγήσω ότι ουδέποτε, ποτέ δεν θα θεωρήσω την αρνητική διάσταση ως μέρος των αρμοδιοτήτων μου. Επεναντίας, όταν ε, λέμε την, ότι υπάρχει ανάγκη να είμαστε παγκόσμιο πρωταθλητές ισότητας, ε, ισότητας των φύλων, κλίματος, μα είμαστε ήδη, ξέρετε, ήδη είμαστε παγκόσμιο πρωταθλητές σε όλους αυτούς τους τομείς. Οπότε καλό θα ήταν να το αποδεχτούμε και με κάποια υπερηφάνεια και να το υπερασπιστούμε. Τώρα αυτό που μου ζητάτε προσωπικώς, αυτό που μου ζητάτε να κάνω είναι ότι τα, να σας, θα σας απαντήσω ότι τα τελευταία 30 χρόνια χτίζω γέφυρες επικοινωνίας και αυτό ήταν η δουλειά μου για να ε, μπορέσουν οι άνθρωποι να βρεθούν κοντά και θα συνεχίσω να το πράττω. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η πράσινη. Ένα λεπτό ο κύριος ε, Ματζίγκ. Κύριε Σχοινά, ξέρω ότι θέλησατε να παρουσιάσετε με θετικό τρόπο τον τίτλο σας, αλλά δεν ε, σας δημιουργεί αμηχανία αυτός ο τίτλος, να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Κοιτάξτε, εδώ ε, από τη δεκαετία του 1990 στο ίντερνετ, πολλοί το θεωρούν αυτό πολύ διαφορετικά. Εμείς θέλουμε ακριβώς να μην έχετε έναν τίτλο που είναι δώρο στους ε, Άρα ανησυχώ ποιε θα είναι για τις προτεραιότητες για την ένταξη. Δεσμεύεστε ότι θα αξιολογήσετε το σχέδιο δράσης του 2016 για τους ε, υπηκόους τρίτων χωρών που ζουν στην Ένωση και ότι θα αποσπάσετε περισσότερου πόρου στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα δεσμεύεστε να στηρίξετε την άμεση χορήγηση πόρων για τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ και την κοινωνία των πολιτών και τι οργανώσει τη για την ένταξη και τι συμφωνίε και τι δραστηριότητε υποδοχή όπω πρότεινε το Κοινοβούλιο στη θέση του για το σύστημα ασύλου. Δύο λεπτά κύριε Σχοινά. Κύριε Ματζίτ, μα νομίζω ότι απάντησα και στην κυρία Ζίπελ προηγουμένως λέγοντας ότι οι εξτρεμιστές και οι λαϊκιστές πρέπει να φοβούνται τις αξίες μας. Όχι αντίστροφα. Και απορρίπτω, τουλάχιστον όσο με αφορά, ο τρόπος που αντιμετωπίζω αυτόν τον τίτλο, απορρίπτω αυτή την εκτίμηση που κάνετε ότι ο τίτλος αυτός έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Για το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας, Απαντώ κατηγορηματικά ναι. Όπω είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία, έχω το πρόγραμμα δράση του 2016, τότε ακριβώ που ήταν η όξυνση τη ε, μεταναστευτική κρίση. Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε διάφορου πόρου από διάφορα τμήματα του προπολογισμού τη Επιτροπή για να έχουμε ένα πρώτο πρόγραμμα δράση για την ένταξη των ε, μεταναστών και προσφύγων. Λειτουργήσε. Αλλά είναι μόνο η αρχή. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Και Είμαστε τυχεροί γιατί οι νέε προτάσει για το πολιτέ δημοσιογών πλαίσιο περιλαμβάνουν τη μακροπρόθεσμη ένταξη των προσφύγων που θα είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Άρα περισσότεροι πόροι, περισσότερε δυνατότητε. Και επίση, σε κάτι άλλο συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Ήσασταν δήμαρχο, έτσι δεν είναι. Στο Σέφιλντ, έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω ότι η εργασία αυτή πρέπει να γίνει στι Βρυξέλλε. Θα ήταν τεράστιο λάθος να θεωρήσουμε ότι οι Βρυξέλλες ε, τα ξέρουν όλα καλά. Όχι, δεν είναι από πάνω προς τα κάτω. Δεν θα σας πούμε τι να κάνετε. Πρέπει να ακούσουμε τις τοπικές κοινωνίες, τις περιφέρειες, τους δήμους, τα άτομα επιτόπου, την κοινωνία των πολιτών και δεσμεύομαι ότι θα με δείτε πολύ. Θα με δείτε στα κέντρα ε, κατάρτισης. Ε, θα με δείτε να παρακολουθώ ποδοσφαιρικά μας στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Θα με δείτε σε όλες τις τοπικές κοινωνίες και βασίζομαι πολύ στη στήριξή σας. Παρακαλώ κύριε Ματζίν, ένα λεπτό. Κύριε Σχοινά, μα κανείς ε, δεν αμφισβητεί πόσο έχετε βλέψει. αλλά με κάθε σεβασμό. Αλλά δεν αρκεί αυτό που είπατε. Όπως είπατε κι εσείς, οι τίτλοι έχουν βάρος και έννοια. Να επιμένετε σε αυτόν τον τίτλο είναι απόλυτη αλαζονία και πολιτική οπισθοδρόμηση, σκοταδισμός για μένα και πολλούς άλλους. Ο τίτλος αυτός είναι απαράδεκτος, απλά και μόνο. Και είναι μία παραχώρηση στους ακροδεξιούς ρατσιστέ και φασιστές. Και μόνο μέσω εγγύηση επαρκού στήριξη και ισχυρή νομική θέση μπορούμε να εγγυηθούμε την ένταξη όλων. Είτε είναι ετούντε άσυλο, μετανάστες ή πρόσφυγες. Επίσης υπάρχουν πολίτες τρίτων χωρών που μένουν πολλά χρόνια στην Ένωσή μας και που παρεμποδίζονται να βρουν δουλειά λόγω των κανόνων. Θα βοηθήσετε την ελεύθερη κυκλοφορία, τροποποιώντας ε, την οδηγία για τους ε, κατοίκους που έχουν μείνει πολλά χρόνια στην Ένωσή μας. Ένα λεπτό κύριε Σχοινά. Δεν είπατε τελικό μου λεπτό. Όχι, όχι, όχι. Τελικό λεπτό για αυτή τη συζήτηση. Γιατί για κάθε βουλευτή έχουμε πέντε λεπτά. Γιατί έτσι που το είπατε, τελικό λεπτό, τελευταίο λεπτό, ακούστηκε λίγο απειλητικό, κύριε Ματζή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω περισσότερο για το πρώτο τμήμα τη ερώτησή σα. Ξέρετε πολύ καλά την στάση μου. Για το δεύτερο τμήμα. Συμφωνώ απολύτω. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να αναθεωρήσουμε την νομοθεσία μας για όσους ε, διαμένουν εδώ και πολύ καιρό στην Ένωσή μας από τρίτες χώρες και προβλέπεται αναθεώρηση. Και μερικές από τις ε, πρώτες αναθεωρήσεις νομοθετημάτων σε αυτόν τον τομέα αποδεικνύουν ότι υπάρχουν κενά και αντιφάσεις σε αυτή την νομοθεσία. Και βεβαίως είμαι διατεθειμένος να εξετάσω την τροποποίηση της νομοθεσίας για τους μακροχρόνια εγκατεστημένους στην Ένωση από τρίτες χώρες για να αρθούν όποια εμπόδια τους εμποδίζουν να ε, επωφεληθούν από την ε, κινητικότητα εργασίας παντού στην Ένωση. Ξέρω ότι αυτό είναι πολύ κοντά στην συνάδελφο που κάθεται δίπλα σας εκεί. Περνάμε στην πολιτική ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ο Νίκολας Μπέι. Ένα λεπτό. Ο προκάτοχός σας, ο κύριος Αβραμόπουλος, θέλησε να φέρει σε αντίθεση με την νόμη με την παράνομη μετανάστευση, την οποία ήθελε να πολεμήσει χωρίς να έχει τα, μέσα. Όλοι ε, μιλάμε για το δικαίωμα του ασύλου, όμως ε, τώρα πια το άσυλο έχει γίνει ένα κομμάτι της μετανάστευσης και οι ετώντες σε άσυλο ε, δεν επαναπατρίζονται ακόμα και όταν η αίτησή τους απορρίπτεται. Οπότε η ελευθερία ε, κυκλοφορίας, αυτό το μεγάλο ιδεώδες, έχει γίνει ε, ελευθερία εγκατάστασης. Είμαι εισηγητής ομάδας μου για την επόμενη οδηγία επιστροφής. Ε, στα, στις 10 σελίδες ε, απάντησή σας ε, στις ερωτήσεις μας δεν αναφερθήκατε καμία φορά σε αυτό. Εσείς έχετε την ευθύνη να προστατεύετε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής ποια είναι τα τεχνικά και νομικά μέτρα τα οποία θα λάβετε προκειμένου να γίνονται οι ε, επιστροφές και τι θα κάνετε έτσι ώστε οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες να λάβουν μέτρα για να την εμποδίσουν την μετανάστευση. Ευχαριστώ. Ο λόγος για δύο λεπτά στον κύριο Σχοινά. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη, ιδιαίτερα όταν μιλούμε για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, είναι μια σχετική τάση να αναζητούμε μία τμηματική, μερική αλήθεια για να εξηγήσουμε το σύνολο του προβλήματος. Δυστυχώς όμως αυτό το πρόβλημα δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε μέσω μιας μερική αλήθεια. Χρειάζεται λοιπόν να τα ξαναδούμε όλα από το μηδέν. Και όπω ε, είπα και στην κυρία Μετσόλα, ότι ο όρος σύμφωνο είναι πολύ ωραίος αλλά χρειάζεται και περιεχόμενο. Έτσι θέλω να πω και σε εσά ότι χρειάζεται να ξαναδούμε όλα τα δεδομένα. Για να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα επιστροφής, χρειάζεται να έχουμε ένα σύστημα συμφωνιών επανεισδοχής με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Και σκοπεύω μαζί με την ε, επίτροπο που είναι υπεύθυνη για τις ε, διεθνείς εταιρικέ σχέσεις ε, με τους άλλους αντιπροέδρους και κυρίως με τον Επίτροπο Διεύρυνσης και Γειτονίας θέλουν να οργανώσουμε ένα τέτοιο σύστημα. Πρέπει να συζητήσουμε με τις τρίτες χώρες και να αναζητήσουμε όχι την ερεσιμότητα Χρειάζεται να αναζητήσουμε σφαιρικές συμφωνίες που θα είναι προς κοινό όφελος. Σε αυτές τις συμφωνίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα αίτια του προβλήματος και τις ανάγκες ανάπτυξης των τρίτων χωρών, να δώσουμε δηλαδή ευκαιρίες στους νέους εκεί να μείνουν στη χώρα τους, αντί να πέφτουν στη θάλασσα και να προσπαθήσουν να ε, κολυμπήσουν, να πέφτουν στα χέρια των κυκλωμάτων διακινητών. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, αυτή είναι η πρόθεσή μου, το έχω συζητήσει με την Ιλβα Γιώχανσον και αυτό μας ζητάει και η ε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι έτσι θα έχουμε καλύτερη, καλύτερες πιθανότητες να πετύχουμε. Ευχαριστούμε. Ο, ακόμα ένα λεπτό στον κύριο Μπέι. Με ανησυχία απάντησή σας δεν φαίνεται πολύ διαφορετική από αυτήν του κύριου Αβραμόπουλου και των προηγούμενων που απέτυχαν. Θέλω να σας ρωτήσω το εξή τώρα. Για τα κυκλώματα διακινητών που περνούν ανθρώπους από την Αφρική στην Ευρώπη σε άθλιες συνθήκες. Υπάρχουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις που είναι συνένοχες. Τι θα κάνετε μαζί με την Frontex έτσι ώστε αυτές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να πάψουν ε, να ε, είναι συναυτουργοί και να πάψουν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους άθλιες μεθόδους. Η, η κυρία Καρόλα Ρακέτε ε, ακούστηκε σήμερα ε, από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ παρόλο που συμμετέχει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ο κύριος Χινάς, δεν συμφωνώ με αυτό το επιχείρημα. Δεν πιστεύω ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι το πρόβλημα που δημιουργεί αυτό το φαινόμενο. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει θα πρέπει να είναι τμήμα τη λύση που θα αναζητήσουμε. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο σφαιρικό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα χωρίς να έχουμε την εξυπνάδα, την ευφυΐα να αντιμετωπίσουμε τις αιτίε του. Είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι είναι θέμα διακινητών, ότι η αιτία, η αιτία είναι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Δεν είναι τόσο απλό τα πράγματα. Το φαινόμενο είναι πολύ πιο περίπλοκο, είναι παγκόσμιο, δεν εξηγείται με απλούς όρους, δεν εξηγείται με κατακαιρματισμό. Σας εξήγησα ότι ο μόνος τρόπος και το μόνο μέσο που έχουμε είναι να κοιτάξουμε λίγο προς τα πίσω, στο παρελθόν, να δούμε τι δεν λειτουργήσε. Και εκεί έχετε δίκιο. Οι επιστροφές δεν λειτουργήσαν. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω και δεν λειτουργήσαν ακριβώς διότι δεν έχουμε αρκετές συμφωνίες επανεισδοχής για να στηρίξουμε αυτή την πολιτική επιστροφών. Οπότε κάτι έμαθα κι εγώ, κάτι έχω μάθει, ότι στην μεταναστευτική πολιτική όλα συνδέονται με όλα τα υπόλοιπα. Now Και πάλι ευχαριστούμε. Και τώρα περνάμε στους εταιρικούς μεταρρυθμιστές, ο κύριος Προκατσίνη. Καλησπέρα σας κύριε Σκηνά. Βλέπετε ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι αποτέλεσμα πολιτισμού και αξιών που μας καθορίζουν ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτική πολυφωνία, διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας, σεβασμός για τις μειονότητες, για τα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων. Για να δώσω μερικά μόνο παραδείγματα. Ποιε συγκεκριμένε δράσει μπορείτε εσεί να, κάνετε και να αποφύγουμε μια κουλτούρα γκαιτοποίηση. Ακριβώ το αντίθετο τη κουλτούρα που θα έπρεπε να μα χαρακτηρίζει, του πολιτισμού που θα μπορούσε να μα χαρακτηρίζει. Μιλάω για γειτονιέ πράστια τη πόλη μα, όπου ιδιαίτερε πολιτιστικέ και θρησκευτικέ ταυτότητε εξαιρούν, αποκλείουν την ευρωπαϊκή κληρονομιά και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Εκεί όπου που ριζοσπαστικές θρησκευτικέ απόψεις που έχουν προκαλέσει πολλές φορές οδύνη και στα κάτι μελη βρίσκουν την ευκαιρία να ανθίσουν. Για δύο λεπτά, κύριε Σχοινά. Κύριε Προκατσίνη, ουδέποτε στη ζωή μου υπερασπίστηκα ή μου άρεσαν ή ε, πρόθεσα έννοιες που τελείωναν σε «ισμός» και νομίζω ότι τα φαινόμενα που ε, αναφέρατε είναι το αποτέλεσμα πολλών τέτοιων ισμών. Και πάλι όμως, τα γκέτο αυτά, εγώ προτιμώ να τα αποκαλώ νήσους αποκλεισμού. Ε, είναι αποτέλεσμα πολυπαραγοντικών εξελίξεων στην κοινωνία. Δεν υπάρχει μία εξήγηση, δεν υπάρχει μία παράμετρος. Μπορώ να σκεφτώ κάμποσες, αλλά δεν υπάρχει μία και μόνο. Ε, κατά τη δική μου την άποψη, η απάντηση για το τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ απλή. Το είπε και στον κύριο Μάντζετ προηγουμένως. Θα πρέπει να ακούσουμε τις πόλεις, τις τοπικές αρχές. Θα πρέπει να πάμε επιτόπου θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ένταξη και συμμετοχή όλων. Πώς θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω προς την κοινωνία μας. Έτσι μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους ισμούς και τις ακραίες ιδεολογίες. Και πάλι εσείς κύριε Προκατσίνη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Σχοινά, στη γραπτή σας απάντηση λέτε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την νόμιμη μετανάστευση και ότι θα είναι ένας από τους κύριους στόχους σας. Συμμερίζεστε την άποψη ότι ο μόνος τρόπος να καθορίσουμε ένα περιφερειακό νόμιμο πλαίσιο για τη μετανάστευση είναι να καταπολεμήσουμε τη λάθρο μετανάστευση. Να πω ότι πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί την πρόθεσή σας να βάλετε τον άνθρωπο, το ανθρωπινό, στο επίκεντρο της πολιτικής σας δράσης. Σε αντιδιαστολή με αυτό που συνήθως συμβαίνει εδώ στο σώμα αυτό, και που συχνά είναι δέσμιο ιδεολογικών προσεγγίσεων. Η δική σας στάση μου θυμίζουν τα λόγια του Ζαν του καθολικού φιλοσόφου, ότι ένα τρισεκατομμύριο ιδέες δεν έχουν την ίδια αξία με ένα ανθρώπινο «ον». Τον άνθρωπο πρέπει να αγαπάμε, γι' αυτόν θα πρέπει να ζούμε και να πεθαίνουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Σχοινά. Είχατε χρησιμοποιήσει μόνο ένα λεπτό στην πρώτη σας απάντηση, οπότε τώρα έχετε δύο. Ευχαριστώ. Κύριε Προκατσίνη, οτιδήποτε θα μας κάνει να βρούμε κοινό έδαφος στο επίπεδο του ανθρωπισμού, ευχαρίστως να πάμε προς τα εκεί μαζί. Ό,τι είναι ανθρωποκεντρικό, εκεί θα βρεθούμε στην ίδια κατεύθυνση και μπορούμε να συμβαδίσουμε για την νόμιμη μετανάστευση. Τρεις λόγοι μας αναγκάζουν να κάνουμε κάτι το ουσιαστικό για την νόμιμη μετανάστευση και είναι και τρεις κέρια σημασία. Πρώτον, γιατί είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις δημογραφικές μας δυσκολίες. Δεύτερον, διότι αυτός είναι ένας τρόπος να διακόψουμε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο των λάθροδιακινητών. Και το τρίτον είναι ίσως ένας από τους πιθανούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε και τις ελλείψεις που έχουμε σε δεξιότητες. Το να κινηθούμε λοιπόν προ μια ουσιαστική λύση για την νόμιμη μετανάστευση δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με την καταπολέμηση τη λάθρο μετανάστευση. Είναι κάτι που πρέπει να διοργανωθεί σωστά, με θετικό τρόπο. Και έχουμε νομίζω κάνει μια καλή αρχή. Τα πιλωτικά προγράμματα που επιτρέπουν σε κάποια από τα κράτη-μέλη μα, με τη βοήθειά μα, να αρχίσουν να ε, εργάζονται και να εφαρμόζουν προγράμματα για την νόμιμη μετανάστευση. Είναι μια καλή αρχή. Πρέπει να κάνουμε όμω και περισσότερα. Και έτσι κι αλλιώς είμαι νέος αυτά τα καθήκοντα, να ξαναδούμε την πρότασή μα για τη γαλάζια κάρτα ενδεχομένω. Ίσως να έχουμε μια προσέγγιση με υπερβολική και ε, απαιτήσει. Να είμαστε ίσως λίγο πιο ε, συμμαζεμένοι στις απαιτήσει μας. Ε, για τους νόμιμους διαδρόμους σε συνδυασμό με την, με την κατάσταση. Και αυτό είναι ένας άλλος εναλλακτικός τρόπος να φέρουμε κόσμο νόμιμα στην Ευρώπη κόσμο που μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη και την άνθηση των κοινωνιών και οικονομιών μας. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στην Ενωτική Ευρωπαϊκή Αριστερά. Ο κύριος Αρβανίτης. Παρακαλώ. Εκπρόσωπος της ΓΚΟΕ, ένα λεπτό. Αξιότιμε κύριε Σκινά, καλώς ήρθατε. σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Χρησιμοποίησατε πολλές φορές τη λέξη ασφάλεια, ασφάλεια, ασφάλεια και σήμερα και χάρηκα πρέπει να σα πω τη λέξη υγεία, υγεία, υγεία και φαντάζομαι ότι θεωρείτε ότι μιλάτε για πρόσβαση όλων των ανθρώπων στην υγεία. Σημαίνει δηλαδή για μένα ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα είδηση εδώ. Διευκρινίστε το αυτό, αν μιλάτε γι' αυτό ακριβώς. Όμως, κύριε Σχοινά, τέσσερις πολιτικές ομάδες, το Renew, οι Σοσιαλιστές, οι Πράσινοι και εμείς οι Γκουε, εμένουμε στο θέμα του τίτλου. Είστε πολύ έμπειρος και απορώ πώς δεν μας καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε το μισό κοινοβουλίο. Ο τίτλο του χαρτοφυλακίου σα για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωή έχει γίνει εργαλείο στην ακροδεξιά. Κυρία Λεπέν πανηγύρισε γι' αυτό. Το ακούσατε κι εσεί. Και πραγματικά θέλω να πω ότι περίμενα από εσά άλλη κίνηση. Μία δήλωση. Δεσμεύεστε λοιπόν να τον αλλάξετε. Είμαι δημοσιογράφος και θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις σε, σε ένα πολύ έμπειρο και αξιόλογο άνθρωπο. Από έναν πολύ έμπειρο και αξιόλογο άνθρωπο. Δεσμεύεστε να τον αλλάξετε όχι μόνο για συμβολικούς λόγους, κύριε Σχοινά, αλλά κυρίως για να μας πείσετε ότι απέχετε από αυτή τη ρητορική που θέλει να διχάσει την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ, κύριε Αρβανίτη. Ε, ναι, για, το, για την πρώτη ε, ερώτησή σας, όντως, κομμάτι των αρμοδιοτήτων μου είναι ειδικά κάτω από την ισότητα και την ισότιμη πρόσβαση όλων στις καθολικές υπηρεσίες υγείας ε, και πνευδίας είναι ακριβώς να βεβαιωθούμε ότι οι πιο ευαίσθητοι, οι πιο ευάλωτοι και οι πιο αδύναμοι δεν θα αποκοπούν από την πρόσβαση, την ισότιμη πρόσβαση σε αυτές τις βασικές υπηρεσίες. Να, κάτι που μας κάνει Ευρωπαίους. Να, κάτι που πρέπει να προστατεύσουμε στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Να, κάτι που πρέπει να δούμε θετικά, όχι αρνητικά. Τώρα μου λέτε ότι η κυρία Λεπέν πανηγυρίζει. Η κυρία Λεπέν δεν πανηγυρίζει. Η κυρία Λεπέν προσπαθεί να εργαλειοποιήσει αυτή τη συζήτηση προς όφελός της. Και περιμένει να δούμε αν εμείς θα τσιμπήσουμε. Αν τσιμπάμε, παίζουμε το παιχνίδι της κυρίας Λεπέν. Αν δεν τσιμπάμε, η κυρία Λεπέν απειλείται από τις αρχές μας. Αυτή είναι η δική μου λογική. Αυτή είναι η δική μου λογική. Δεν τον αλλάζετε λοιπόν, οπότε είναι ιδεολογικό. Oh, <laughs> συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν σα έδωσα το λόγο. Περίμενα ε, να δω αν έχει τελειώσει ο κύριο Χινά. Γιατί δεν ε, εξήγησε το χρόνο του. Έχετε και μερικά δευτερόλεπτα. Ναι, είχα ένα συνολικό επιχείρημα, μπορώ να το κάνω. Όταν ήρθα εδώ, η ομάδα μου μου ε, είπε Πες ό,τι θες, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά ένα πράγμα μην κάνεις. Μην αντιμετωπίσεις τους ευρωβουλευτές ως δημοσιογράφους. Μην το κάνεις αυτό. Και πραγματικά δεν το έκανα. Αλλά δεν περίμενα ένας ευρωβουλευτής, αντί να μου μιλήσει ως ευρωβουλευτής, να μου μιλάει ως, δημοσιογράφος. Αυτό ομολογουμένως δεν το περίμενα. Και τώρα παρακαλώ, αυτό το λόγο κύριε Η Τιμή μου που είμαι δημοσιογράφο και υπερασπίστηκα τα δημόσια στο δημόσιο σφαίρο, κύριε Σχοινά. Ελπίζω και εσεί από τη θέση σα να κάνετε το ίδιο για του φτωχού, για του ανθρώπου που έχουν ανάγκη. Επιμένω όμω. Στο χαρτοφυλάκιό όσα η ασφάλεια συνδέεται με το μεταναστευτικό σε μια ανησυχητική υπερσυγκέντρωση εξουσιών και την αυθαίρετη σύνδεση τη προστασία των πολιτών με τη θωράξη των συνόρων. Αντίθετα, απουσιάζει εντυπωσιακά μια λέξη, κύριε Σχοινά. Η λέξη δικαιοσύνη. Ρωτώ λοιπόν, δέχεστε να παληφθεί η ασφάλεια από το χαρτοφυλάκιό σα ω ασύμφωνη με τον πραγματικό χαρακτήρα του καθηκόντων σα. Δέχεστε τη λέξη και την ουσία δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Thank you. Now, Mr. Skinas, you... Το τελευταίο λεπτό αυτού του πρώτου γύρου ερωτήσεων, του πρώτου γύρου των συντονιστών. Παρακαλώ. Κύριε Βανίτη, σέβομαι απόλυτα την δικαιοσύνη έτσι όπως την εννοείται. Η μόνη διαφορά είναι ότι η δικαιοσύνη δεν είναι στην Αντιπροεδρία τη δικιά μου, δεν είναι στις εντολές που έχω λάβει από την εκλεγήσα πρόεδρο. Είναι η συνάδελφός μου η κυρία ε, Γιούροβα που θα δείτε ε, τη Δευτέρα εδώ και θα σας εξηγήσει. Τώρα μου λέτε αν δέχομαι να βγάλω την ασφάλεια, αντιλαμβάνομαι καλά, από το χαρτοφυλάκιό μου. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η ασφάλεια και η μετανάστευση και η πολιτική μετανάστευση ε, σχεδόν σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μαζί. Στην Ελλάδα, τη χώρα που και οι δυο ξέρουμε καλά, είναι μαζί. Σε πολλές άλλες χώρες είναι μαζί. Ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ θα σας πει ότι και στη Λίμπε είναι μαζί. Και στην Κομισιόν Γιούγκερ επίσης ήταν μαζί. Με αντιπρόεδρο τον κύριο Τίμερμανς και επίτροπο τον κύριο Αβραμόπουλο, ώσπου να έρθει ο κύριος Κίνγκ. Γιατί λοιπόν στην Κομισιόν Φαντερ Λάινεν να είναι διαφορετικά, λέω εγώ. Σε κάθε περίπτωση η λογική είναι δεδομένη, είναι μέσα σε ένα πλαίσιο αποφάσεων που σύμφωνα με τη συνθήκη είναι το άρθρο 17 σημείο 6 της συνθήκης που δίνει στον πρόεδρο της Επιτροπής την απόλυτη αρμοδιότητα νομική, θεσμική, να χτίσει την Επιτροπή όπως θέλει, ακούγοντας βέβαια και ε, διαλέγοντας με εσά και λαμβάνοντας ψήφο εμπιστοσύνη όπως έλαβε τον Ιούλιο. Άρα ε, το λέω αυτό για να σας πω ότι δεν εξαρτάται από μένα εδώ να πω έτσι κι αλλιώ, αλλά μπορώ κάλλιστα για να απαντήσω στην ερώτησή σας να σας θυμίσω ποια είναι η κατάσταση η ισχύουσα, η τρέχουσα. Και η κατάσταση η τρέχουσα είναι απολύτως η ίδια με αυτή τη δικιά μας, την τωρινή. Ευχαριστώ. Ανά και τώρα να δώσω το λόγο στην συμπρόεδρο κυρία Φερχάιν. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Και σας ε, υπενθυμίζω ότι πρέπει να τηρούμε το χρόνο μας, γιατί ήδη έχουμε καθυστέρηση. Πρώτα απ' όλα από την Επιτροπή Πολιτισμού και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Τόμας Φραντχόφσκι. Ως αντιπρόεδρος θα είστε υπεύθυνο για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον αθλητισμό. Να σας ρωτήσω κάτι για τον αθλητισμό. Μία από τις πιο επιτυχείς πρωτοβουλίες της προηγούμενης Επιτροπής ήταν η συνεργασία τρίων επιτρόπων υγείας, αθλητισμού και πολιτισμού ούτω ώστε να βελτιώσουμε την υγεία των συμπολιτών μας. Και άλλο καλό παράδειγμα για τον αθλητισμό είναι η διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Προτίθεστε να συνεχίσετε αυτές τις πρωτοβουλίες και αν ναι, πώς θα τις βελτιώσετε. Πώς θα συνεχίσετε λοιπόν αυτές τις καλές πρωτοβουλίες που ήδη υπάρχουν. Ευχαριστώ κύριε Φρανκόφσκι. Κύριε Σχοινά, παρακαλώ δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φρανκόφσκι. Ναι. Οι πρωτοβουλίες αυτές, αυτού του είδους πρωτοβουλίες, είναι καλύτερες. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία. Γιατί είναι πρωτοβουλίες ε, μεγάλης ε, κλίμακας, διαμεθοριακές, που αγγίζουν πολλούς συμπολίτε. Έτσι αυξάνεται η ευαισθητοποίηση και η κατανόηση του τι μας ενώνει. Και αναμφίβολα, ο αθλητισμός μας ενώνει. Το ίδιο ισχύει και για την υγεία. Ένας υγιεινός, υγιής τρόπος ζωής έχει να κάνει πολύ με τον αθλητισμό. Και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την ε, Κυπρία συναδελφό μου, την κυρία Στέλλα Κυριακίδου. Θέλω να αξιοποιήσω πλήρε τι δυνατότητε συνεργασία ε, μεταξύ τη κυρία Γκάμπριελ, τη κυρία Κυριακίδου. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο που δεν αναφέρατε. Και είμαι στον πειρασμό να το αναφέρω και αυτό για να ολοκληρώσουμε την εικόνα. Ο αθλητισμό είναι και ένα θαυμάσιο δρόμο για να ενταχθούν πολλοί συμπολίτε μα στι κοινωνίες μα, όπω είπε ο κ. Ματζίντ, με τέτοιες πρωτοβουλίες καταλαβαίνουμε όλοι ότι ανήκουμε στην ίδια κοινωνία. Έτσι έχουμε πιο ανθεκτικές κοινωνίες, με περισσότερη κοινωνική συνοχή. Και προετοιμαζόμενος για τη συζήτησή μας, με ενθουσιασμό είδα ότι εδώ κοντά, όχι πολύ μακριά, στο Κράινεμ υπάρχει ο ποδοσφαιρικός εραστρανικός ε, όμιλος ε, του Κράινεμ. Με τη βοήθειά μας μέσω του έρασμου ΣΥΝ, χρηματοδότηση δηλαδή από εκεί, κατάφεραν να εντάξουν πολλούς ε, μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι ένα πρόγραμμα καταπληκτικό που θα επισκεφθώ τάχιστα. Αυτού του είδους πρωτοβουλία εκ των κάτω στον αθλητισμό μπορούν να βοηθήσουν, πρωτοβουλίες μπορούν να βοηθήσουν. Εδώ πρέπει να δώσουμε πόρους, εδώ πρέπει να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Φρανκόφσκι. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ναι, μα πήγα στο Κράινεμ ακριβώ. Είμαι νέο μέλο τη Επιτροπή Πολιτισμού. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που είπατε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση ε, ανέβηξε πολλέ καλέ πρωτοβουλίε. Για παράδειγμα, έχουμε διάφορα κύπελα αθλητικά. Επίση, ε, διάφορα πιλωτικά προγράμματα για την ένταξη προσφύγων. Θα συνεχίσετε αυτές τις πρωτοβουλίες και πώς θα τις βελτιώσετε, πώς θα τις ε, ενισχύσετε. Κύριε Σχοινά, παρακαλώ. Όπως είπα προηγουμένως για τα θέματα μεταναστών και προσφύγων, θα ξαναδούμε το σχέδιο δράση του 2016 για την ένταξη των μεταναστών και προσφύγων. Και πρέπει να γίνει αυτό. Για ένα πολύ απλό λόγο. Όταν ε, το εκπονήσαμε ήμασταν στο 2016. Ήταν τη στιγμή όπου να μην γελιόμαστε. Η αντίδραση της Ένωσης ε, στις μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυσμών στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μας ανάγκασε να ασχοληθούμε περισσότερο με την διαχείριση του προσφυγικού φαινομένου δεν είχαμε ακόμη την τεχνογνωσία και τους πόρους να ασχοληθούμε περισσότερο με την ένταξη. Αλλά παρά τις δυσχέρειες, οι υπηρεσίες μας, ε, η Γενική Διεύθυνση Home, αλλά και οι άλλες υπηρεσίες που συνεργάστηκαν, όλοι αυτοί λοιπόν εκπώνησαν αυτό το πρόγραμμα δράση. Τώρα πρέπει να το αναθεωρήσουμε. Τώρα ακριβώ είναι στιγμή να το αναθεωρήσουμε για να κάνουμε περισσότερα. Και μάλλον καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σχοινά. Ε, Επόμενο ομιλητή, ο κ. Μάτικτ από την Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευση. Σοσιαλιστέ. Κύριε Σχοινά, ο πολιτισμός πραγματικά δημιουργεί την αίσθηση του ανήκειν. η γενική εκπαίδευση, η γενική παιδεία μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να ενταχθούν στον κόσμο και στην κοινωνία τους. Ε, πώς οι νέοι λοιπόν θα έχουν καινούριε εμπειρίες, ε, καινούριε ικανότητες ε, και να ενταχθούν στην κοινωνία μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Πώς σκοπεύετε να προωθήσετε την αίσθηση του να ανήκει κάποιος στην Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Κύριε Σχοινά, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Αυτό που μας ορίζει, που μας καθορίζει και μας δίνει την ε, ε, κοινή αίσθηση του ανήκει είναι ακριβώς ο πλούτος και η ποικιλία της κουλτούρας μας και του πολιτισμού μας. Ε, γι' αυτό το λόγο μας θαυμάζουν και θα έλεγα και μας ζηλεύουν σε όλο τον κόσμο. Είναι αρκετό αυτό, όχι δεν είναι, δεν είναι. Αφενός χρειάζεται να συνεχίσουμε να προωθούμε και να επενδύουμε στην πολιτιστική μας ποικιλία και στον πολιτιστικό μας πλούτο και από την άλλη μεριά μέσω της εκπαίδευσης να ε, δημιουργήσουμε ένα πιο ενιαίο αφήγημα. Έχετε δίκιο, μέσω της εκπαίδευσης θα πρέπει να ενώσουμε τους ανθρώπους, να τους φέρουμε κοντά τον ένα στον άλλο, να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ε, περιοχή εκπαίδευσης, ε, ένα ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης, συγγνώμη, και ε, αυτό να αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Χρειαζόμαστε μια κάρτα μαθητή-φοιτητή, χρειαζόμαστε να χτίσουμε τις Ευρωπαϊκές Συμμαχίες Πανεπιστημίων που έχουν ήδη ξεκινήσει. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε ε, και να δώσουμε πιο ισχυρό ρόλο στους εκπαιδευτικούς γιατί κάνουν ένα εξαιρετικό έργο, συνεισφέρουν στις κοινωνίες μας και τέλος θα πρέπει να διαθέτουμε και τα απαραίτητα κονδύλια γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή ε, τα κονδύλια δίδονται μέσω του Ταμείου του Εράσμους ΣΥΝ ε, που ε, είναι τα στολίδια του στέματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε προτείνει να τριπλασιαστούν οι, οι πόροι και βέβαια έχουμε και το Discovery U και το σώμα αλληλεγγύης ε, που είναι πολύ σημαντικές προτεραιότητες επίσης. Επίσης συμφωνώ ότι για το Discovery Europe EU και για το ε, σώμα αλληλεγγύης αυτοί που θα συμμετέχουν δεν θα πρέπει απλώς να ταξιδεύουν, θα πρέπει να επιστρέφουν με εμπειρίες, θα πρέπει να εκτίθενται σε καινούριε δεξιότητες και να φέρνουν πίσω μια γνώση την οποία θα την αποδώσουν στην κοινωνία τους και θα εργαστώ σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση από τον κύριο Μάτιτς. Οι πρόσφατες εκλογές έδειξαν ότι οι νέοι θέλουν να, ε, μια δράση εναντίον της κλιματικής αλλαγής και, της και υπέρ της βιωσιμότητας. Πώς θα επιτρέψετε σε αυτούς τους νέους να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα. Ο κ. Σχοινάς. Χωρίς αμφιβολία, το πράσινο κύμα θα είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ε, καινούριας Κομισιόν. Δεν είναι κάτι μυστικό. Δεν χρειάζεται να μας πείσετε γι' αυτό. Νομίζω ότι είμαστε πεπισμένοι ήδη και είμαι σίγουρος ότι έχετε ακόμα στο μυαλό σας την ομιλία της εκλεγής σας ε, Προέδρου τον Ιούλιο που μίλησε πάρα πολύ για την πράσινη Ευρώπη και βέβαια για την ψηφιακή Ευρώπη ε, μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι πολύ ψηλά. Σίγουρα ένα κομμάτι αυτής της προσπάθειας ε, εξαρτάται από τους νέους, από τη συμμετοχή των νέων, διότι οι νέοι Φέρνουν μια καινούρια οπτική στον αγώνα μας αυτό. Με εξέπληξε που διάβασα μερικές, ε, ε, μερικά άρθρα που προσπαθούν να διδάξουν στους ε, νέους για το πώς πρέπει να εκφράσουν τις απόψεις τους για το κλίμα. Δεν πρέπει να απολογούνται οι νέοι, έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους όπως νομίζουν. Οπότε από την δική μου πλευρά ευθυνών και μέσω των προγραμμάτων που αφορούν τους νέους, το Σώμα Λεγγύης και το Discovery You, θα κάνω ό,τι μπορώ για να προωθήσω τους νέους στον αγώνα για τη βιωσιμότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Θαγάν από την Επιτροπή Πολιτισμού και την Ομάδα ΡΙΝΙΟΥ. Κύριε Σκηνά, ήθελα να συμφωνήσω με την άποψη για τον τίτλο του χαρτοφυλακίου σα. Είτε πρόκειται για μετανάστευση, είτε για πολιτισμό, δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το υψηλότερο μήνυμα και καλό θα να αλλάξει. Όταν μιλάμε τώρα για εκπαίδευση και παιδεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε αυτό θα θέσω την ερώτησή μου, υπάρχουν δύο παράλληλε πραγματικότητε. Μία ε, Ευρώπη η οποία αποκτά γνώσει και μία που βρίσκεται σε τέλμα. Από τι πρόσφατε μελέτε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο ε, πτυχιού δικαιούχων τη εκπαίδευση, εκπαίδευση, με 40% σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και που είναι ε, αυτοί που υποφελούνται περισσότερο από το Erasmus Συν. Και μετά υπάρχει και ένα μεγάλο μερίδιο ε, παιδιών με μεγάλε δυσκολίε. Πραγματικά σήμερα στην Ευρώπη ένα, από τα, ένα στα πέντε παιδιά των 15 ετών βάσει τη Ευρωστάτ δεν μπορεί να γράψει, να κάνει αριθμητικέ πράξει ή να διαβάσει. Και ε, αυτό αφορά και τα παιδιά των μεταναστών και το χαρτοφυλάκιο των αμοδιοτήσεων σα βεβαίω. Για, όνομα λοιπόν τη δικαιοσύνη και τη ισότητα, τη αλληλεγγύη που είναι μέρο τη επιστολή ε, ε, και των αρμοδιοτήτων που σα αναθέτει αυτή, πώ εσεί θα αναλάβετε δράση, πώ θα συνδυάσετε αυτέ τι δύο παράλληλε πραγματικότητε. Κυρία Θαγό, ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι στην, στο κέντρο της ερώτησής σας βρίσκεται το θέμα της ε, ισότητας των ανισοτήτων. Πράγματι, Παρά τις πρόοδους μας, παρά τα βήματα που έχουν γίνει, ανισότητες υπάρχουν ακόμα. Και στην αγορά εργασίας και στην ε, εκπαίδευση. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τις αντιμετωπίσουμε. Ιδίως σε μια στιγμή όπου η Ευρώπη βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ για την απασχόληση. Ακριβώς τώρα πρέπει να χτυπήσουμε ε, στο θέμα των ε, ανισοτήτων. Όπως είπε ο κύριος Γιούνκερ, τώρα πρέπει να επισκευάσουμε τη στέγη, στη λιακάδα όταν ο ήλιος λάμπει. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε τις ανισότητες και από τις δύο οπτικές γωνίες, από την αγορά εργασία και την κοινωνική πολιτική, αυτό που θα γίνει σε συνεργασία με τις σε συνδυασμό με τι πολιτικέ του εξαμήνου και τι συστάσει ένα χώρα που εκδίδονται ετησίω, δουλειά την οποία θα αναλάβει ο συνάδελφο φίλο αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκη και όπου θα συμμετάσχω ένεργα, διότι σκεφτείτε, 60% των συστάσεων που κάνουμε προ τα κράτη-μέλη αφορούν ακριβώ τον τομέα των αρμοδιοτήτων μου. Την πρόσβαση στην υγεία, στις δεξιότητες ε, και σε ό,τι απαιτεί επαγγελματικέ ικανότητες. Ε, στη δουλειά λοιπόν αυτή του Ευρωπαϊκού Ξαμήνου θα αξιοποιήσουμε και άλλα εργαλεία, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τους μηχανισμούς για την επαγγελματική κατάρτιση. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν και καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε. Είναι προτεραιότητά μας ούτως ή άλλως και είναι μια προτεραιότητα η οποία θα λάβει τη δέουσα προσοχή. Ε, το λέω με μεγάλη αισιοδοξία. Ε, και επίση συμμερίζομαι την άποψή σα για το πώ θα πρέπει να έχει δημοκρατικότερο χαρακτήρα το Erasmus Συν. Ε, διότι υπάρχουν κάποιε πτυχέ του Erasmus Συν που ε, δυσκολεύουν κάποιε ομάδε του πληθυσμού να συμμετάσχουν επειδή δεν έχουν τα οικονομικά μέσα. Δεν μπορούν να συμβάλλουν, να πληρώσουν όσα χρειάζονται. για να καλύψουν την όσα λείπουν από την κοινοτική συμβολή. Ο συνάδελφος Νίκολα Σμιτ ε, για την απασχόληση και την εργασία ε, θα είναι συνομιλητής μου για να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε κονδύλια από το κοινωνικό ταμείο και να επιτρέψουμε στους νέους αυτούς να έχουν την χρηματοδότηση που θα τους επιτρέψει μαζί με τη δική μας την ε, χρηματοδότηση να προχωρήσουν. Είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Θαγό, έχετε δεύτερη συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω για την σχέση απασχόλησης και εκπαίδευσης και κάτι άλλο που αναφέρατε στην επιστολή αρμοδιοτήτων σας, για την διαχείριση των δεξιοτήτων. Δηλαδή θα πρέπει λιγάκι να κοιτάξουμε τι θα συμβεί στο μέλλον, να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε, να προλάβουμε. Αυτό είναι και μια δέσμευση που έχουμε λάβει για μια Ευρώπη της καινοτομία, για την πράσινη αυτή αλλαγή πώς ε, και το λέω εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, πώς θα προσαρμόσουμε τις, ε, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, πώς θα κοιτάξουμε να επιτρέπουμε την διαρκή ενημέρωση των δεξιοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου και αυτό ώστε κάποιος να παραμένει πάντοτε ενεργός. Κύριε Σχοινά, στις δεξιότητες πρέπει να πορευτούμε βάσει τριών αρχών Πρώτα απ' όλα η αρχή της, του σκοπίμου του κατά πόσον είναι κάτι πρόσφορο και μετά της συμβατότητας και της συμμετοχής. Πρέπει να έχουμε αυτές τις τρεις αρχές υπόψη όταν προετοιμαζόμαστε για να κάνουμε κάτι για τις δεξιότητες σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία, σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Ε, εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ομολογώ, το θέμα αυτό των δεξιοτήτων ε, είναι κάτι που είναι διασκορπισμένο στις αρμοδιότητες μεταξύ πολλών γενικών διευθύνσεων. Με ακούνε κάποιοι από όσους βρίσκονται παρόντες και στην αίθουσα και δουλεύουν σε αυτές τις γενικές διευθύνσεις. Πρέπει αυτός ο κατακαιρματισμός να πάυσει. Σε πολιτικό επίπεδο, είναι αυτό μια δουλειά που θα αναλάβουμε από τη μια ο κύριο Σμιτ που ασχολείται με τα θέματα των δεξιοτήτων και εγώ ο ίδιος. Ε, και αυτό γιατί πρέπει να βρούμε τρόπο να συνεισφέρουμε με πολύ απτό τρόπο και τα πολιτικά μας εργαλεία. Ό,τι είναι κλασική πολιτική απασχόληση θα το αναλάβει ο κύριος Σμιτ και ο κύριος Ντομπρόφσκης. Αυτή είναι η κατανομή αρμοδιότητα. Και η Μαρία Γκάμπριελ με τη δικά της τα μέσα και εργαλεία θα βρεθεί στο πλευρό μας στο επίπεδο της Αντιπροεδρίας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα διοργανωθούμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόμτς από την Επιτροπή Απασχόλησης και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σχοινά, εδώ είμαι. Θα ήθελα να ασχοληθώ με το θέμα ακριβώς των δεξιοτήτων. Διότι θα είστε υπεύθυνο για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Είναι θέμα της Επιτροπής Απασχόλησης, άρα δικό μας. Θέλουμε να διατηρήσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Άρα πρέπει να λειτουργεί σωστά η αγορά εργασίας. Στην Ένωση είναι υψηλά τα ποσοστά απασχόλησης, αλλά παρόλα αυτά έχουμε λήψεις ε, ειδικευμένου προσωπικού σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς και κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα. Και θα κάνετε αυτό που χρειάζεται για να έχουμε μια νέα πολιτική δεξιοτήτων για την Ευρώπη και για την επαγγελματική κατάρτιση των νέων μας. Τι μέτρα θα προτείνετε προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε τα άτομα να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την οικονομία μας. Ποια είναι τα σχέδιά σας λοιπόν για τον τομέα αυτό. Παρακαλώ. Κύριε Σχοινά, παρακαλώ, δύο λεπτά. Πρώτον, κύριε Τόμτς, χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή Απασχόλησης ε, συμμετέχει σε αυτήν την ακρόαση. το γεγονό ότι δίπλα στην Επιτροπή Ελευθεριών και Πολιτισμού έχουμε και την Επιτροπή Απασχόλησης συμπληρώνει την έννοια της αντιπροεδρίας μου. Ακριβώς, συνδυάζουμε όλους αυτούς τους τομείς πολιτικής. Χαίρομαι λοιπόν που είστε μαζί μας. Τώρα για τις δεξιότητες. Δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε ταυτόχρονα. Πρώτον, όπως έλεγα και στην κυρία Φάγων πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δεξιότητε που είναι κατάλληλε για την αγορά εργασία και για να καταπολεμήσουμε τι ανισότητε. Αυτό είναι, α πούμε, ο παραδοσιακό τρόπο επενδύσεων στην ανάπτυξη δεξιότητων. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που επίση έχει μεγάλη σχέση και εδώ πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Είναι το θέμα των λεγόμενων υπείων δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με το πώ θα μπορέσουν να ενταχθούν κάποια άτομα. Όχι δεξιότητε που θα σου δώσουν δουλειά απευθεία, αλλά δεξιότητε που θα σου επιτρέψουν να ενταχθείς καλύτερα στην κοινωνία που ζεις. Πώς να μιλήσεις με άλλους, ε, να πας σε μουσεία, να συμμετάσχεις σε δραστηριότητες κοινωνίας των πολιτών, να παίξεις μπάλα, ε, να βγεις από τον κέτο σου, όπως είπε ο κ. Προκατσίνη. Και αυτές οι δεξιότητες είναι εξίσου σημαντικέ. Όσο και οι δεξιότητες για να βρεις δουλειά. Και είμαστε διατεθειμένοι με τη βοήθεια τον Σμιτ και Γκάμπριλ να ασχοληθούμε και με τους δύο αυτούς τομεί και μέσω νομοθεσία. υπάρχει η νομοθεσία από αυτών μέσω όλων των μέσων που έχουμε μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Erasmus του, του, του Σώματος και του Discovery EU αλλά και μέσω του Horizon 2020 που έχει πολύ αξιοσημείωτη πρικοδότηση για επενδύσεις σε δεξιότητες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Συλλογματική ερώτηση, κύριε Κυρία Τόμιτς, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση αυτή. Να σας υπενθυμίσω τώρα κάτι άλλο. Η Ένωση δεν αντιμετωπίζει μόνο έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, αλλά και ελλείψεις σε ορισμένες δεξιότητες ε, υψηλού επίπεδου. Για παράδειγμα για την ψηφιοποίηση διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε επαρκείς εργαζόμενους αυτό συμβαίνει τώρα. Δεν είναι κάτι μέλλοντο. Πολλά άτομα ε, έχουν δυσχέρειε προσαρμογή. Δεν είναι όλοι νέοι, δεν μπορούν όλοι να προσαρμοστούν στι ε, μεταβαλλόμενε συνθήκε αγορά εργασία. Δεν είναι όλοι ψηφιακά καταρτισμένοι και κατάλληλοι για να καταρτιστούν. Πολλά άτομα λοιπόν ε, δεν έχουν τι αναγκαίε δεξιότητε για να προσαρμοστούν. Πρέπει και αυτού να μην του ξεχάσουμε στην αγορά εργασία, γιατί είναι ακόμη οι συμπολίτε μα. Τι θα κάνουμε για αυτού. Τι θα κάνουμε για αυτού που δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Έχετε συγκεκριμένα σχέδια για αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό κύριε Σχοινά. Ναι. Και εδώ διτή προσέγγιση. Πρώτον. Πρώτα απ' όλα είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων. Αυτό που λέμε upskilling. Δηλαδή τα τμήματα της κοινωνίας που είναι αποκλεισμένα από κάποιες δεξιότητες μπορεί πραγματικά να ανέβουν στο επίπεδο για να μπορέσουν να αποφεληθούν από την ψηφιακή τεχνολογία. Σωστά εντοπίσατε ηλικιωμένα άτομα και άλλε ευάλωτε ομάδε. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για την κοινωνική πλευρά των αρμοδιοτήτων μου. Η άλλη πλευρά είναι ακριβώ να γεφυρώσουμε το χάσμα δεξιοτήτων, όπω το λέμε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το γεγονό ότι τα επόμενα χρόνια θα χρειαστούμε 250.000 ειδικού για την ψηφιοποίηση. Και δεν του έχουμε. Πού θα του βρούμε. Εδώ θα βοηθήσει και η νόμιμη μετανάστευση. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει θετική παρέμβαση μέσω αυτού που η Μαρία Γκάμπλ σας ε, εξήγησε. Η πράξη, το νομοθέτημα για την ψηφιακή εκπαίδευση. Πώς θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητε για να βρούμε αυτά τα άτομα, να τα καταρτήσουμε. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν παράλληλα. Ευχαριστώ. Ε, Επόμενη στη σειρά η κυρία Ιντζήρ από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, την ομάδα των Σοσιαλιστών. Θα μιλήσω σουηδικά, αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σχοινά. Στι απαντήσει σα, στι γραπτές σας απαντήσεις για την νόμιμη μετανάστευση και την ενσωμάτωση, μιλάτε για το γεγονό ότι οι φυστάμενα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με καλύτερο τρόπο. Δεδομένου ότι η Ursula von der Leyen έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην δημιουργία νόμιμων διαδρόμων μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Ε, θα ε, αναρωτιόμουν αν πράγματι τα υφιστάμενα εργαλεία είναι αρκετά. Δεν ξέρω αν η πρότασή σας θα βελτιώσει πραγματικά την κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη επιτροπή. Δεν θα έχετε καινούριε προτάσεις, δεν ετοιμάζετε καινούριε προτάσεις για την νόμιμη μετανάστευση. Έτσι πρέπει να το ερμηνεύσουμε. Δηλαδή δίνεται έμφαση αποκλειστικά στα πιλωτικά προγράμματα της στήριξη τρίτων ε, χωρών και στα υφιστάμενα εργαλεία. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, μάλιστα, υπάρχουν και επιφυλάξει. Τι θα κάνετε έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι θα υφίστανται νόμιμοι διάδρομοι σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε κανεί να, διακι... να μην διακινδυνεύει τη ζωή του για να ξεφύγει από τον πόλεμο και τη φτώχεια. Ο κ. Κινά έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Εντζήρ. Είναι κρίσιμο αυτό το ερώτημα ε, σε σχέση με όλα όσα συζητούσαμε σήμερα. Νόμη μετανάστευση. Ναι, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας χωρίς πάθος και φόβο, με αντικειμενικό τρόπο. Σας ανέφερα τους τρεις λόγους που μας υποχρεώνουν να το κάνουμε. Η δημογραφία, το να ε, σταματήσουμε να καταργήσουμε το μοντέλο των διακινητών, το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών και η γεφύρωση του χάσματος των δεξιοτήτων. Αυτά είναι τα τρία. Μπορείτε να βάλετε όποιες ταμπέλες θέλετε σε αυτά και μάλιστα κάποιοι μου επιτέθηκαν σε ορισμένες χώρες εξαιτία των γραπτών μου απαντήσεων ακριβώς. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε έτσι, για να είμαστε λίγο πιο ευφυείς σε ό,τι ε, αφορά αυτό το θέμα. Πρώτον, να δούμε τι έχει λειτουργήσει και τα πιλωτικά προγράμματα είναι μια πρώτη ε, ντροπαλή, περιορισμένη προσπάθεια, ένα μικρό βήμα που έχει δείξει ότι λειτουργεί. Και μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Μίλησα και με τη συνάδελφό μου την Ιλβα Γιώχανσον αλλά και με τον Γενικό Διευθυντή έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε ακόμα καλύτερα τα πιλωτικά προγράμματα. Δεύτερον, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την πρότασή μας για την μπλε κάρτα, να δούμε γιατί δεν λειτουργήσε. Ίσως ήταν πιο πολύ περιοριστική, ίσως επειδή δεν ήταν αρκετά προσαρμοσμένη στις ανάγκες ε, κάθε φορά. Θα πρέπει να το ξαναδούμε, εν πάση περιπτώσει. Τέλος, κάτι άλλο συναφές που το αναφέρετε, είναι οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι οι οποίοι θα πρέπει να συνδυάζονται με δεσμεύσεις για επανεγκατάσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την νόμη μετανάστευση, έχει λειτουργήσει τοπικά, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερους διαδρόμους και θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας σε αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Ιντζήρα, έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Μάλιστα. Και πάλι στα Σουηδικά. Δεν νομίζω ότι μου δώσατε κάποια καινούρια απάντηση, κάποιο καινούριο στοιχείο που να αναγγέλει κάποιες ε, καινούριες πρωτοβουλίες, κάτι καινούριο σε σχέση με τα όσα έχουν ήδη δοκιμαστεί. Εν πάση περιπτώσει, στην γραπτή σας απάντηση για την ενσωμάτωση, λέτε ότι οι λύσεις θα πρέπει να έρθουν από κάτω, όχι από την κορυφή, αλλά από τη βάση. Και ε, μιλήσατε για τη σημασία τη ευρωπαϊκή σηματοδότηση. Θα στηρίξετε τι προσπάθειε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε μια ελάχιστη ευρωπαϊκή στήριξη για, την, ε, ε, για το Ταμείο μετανάστευση και ασύλου και ότι θα ενδυναμώσουμε το ρόλο των τοπικών αρχών έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ζητούν χρήματα συνεχώ από τι κεντρικέ κυβερνήσει, αλλά να μπορούν να χρηματοδοτηθούν κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχουν κάποιε κεντρικέ κυβερνήσει που ε, δεν θα, το, ε, δεν θα ε, επέτρεπαν αυτή τη χρηματοδότηση. Ε, είμαι αντιπρόεδρο ομάδα ποικιλομορφία και μειονοτήτων Πώς θα υποστηρίξετε τις μειονότητες στην Ευρώπη, γιατί η ακροδεξιά ενισχύεται όλο και περισσότερο. Και ο έχει ένα λεπτό. Πολλές ερωτήσεις για ένα λεπτό, θα προσπαθήσω. Για το ταμείο, για, τα, για, τα, για τους πόρους, για τα κονδύλια. Ε, ε ήρθα σε πολλές επαφές ε, ε, πριν έρθω εδώ με πολλούς ανθρώπους και ε, δεν είδα, δεν ένιωσα ότι η πρικοδότηση του Ταμείου Ασύλου και είναι μικρή. Ε, έχουμε φτάσει από τα 10 στα 30 δισεκατομμύρια ε, για αυτές τις πολιτικές. Τριπλασιασμό δηλαδή. Τώρα μου λέτε ότι θα πρέπει να δεσμευθώ ένα κομμάτι από αυτά τα ποσά να πηγαίνει κατευθείαν σε τοπικές και περιφερειακές αρχές. Λυπάμαι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, διότι εσείς είστε οι συνομοθέτε. εσείς αποφασίζετε το περιεχόμενο των νομοθετικών μας κυμάτων. Αν λοιπόν εσεί πείσετε το Συμβούλιο θα σας στηρίξω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η ε, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να έρθουμε με άλλο τρόπο σε επαφή με τις τοπικές αρχές τώρα. Ε, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μου δει περισσότερο χρόνο για να μιλήσω και για τις μειονότητες που με ρωτήσατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολλές ερωτήσεις για ένα λεπτό, αλλά πρέπει να τηρούμε τον χρόνο. Και τώρα, κύριος Μπρόια, από την Επιτροπή Λίμπε, πράσινη. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε σκηνά όπως, ε, πολιτικές όπως το Μητρό Επιβατών. Οι πολιτικές όπως η τήρηση των δεδομένων ε, και το Μητρό ε, Επιβατών. Η καταγραφή των ιδιωτικών επικοινωνιών και των καθημερινών μετακινήσεων. Αυτό κάνει τους πολίτες να αισθάνονται διαρκώς ότι παρακολουθούνται, ότι υποκλέπτονται οι επικοινωνίες τους. Ε, δεν ε, αισθάνονται ότι είναι ελεύθεροι και ότι μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και μια ίση κοινωνία. Ε, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δις κατέληξε στην απόφαση ότι οι πολίτες που σε καμία περίπτωση δεν έχουν την παραμικρή σχέση με εγκληματική οργάνωση περιλαμβάνονται σε αρχή όπως το PNR και τηρούνται τα στοιχεία τους για πολύ καιρό. Δεν έχουν λοιπόν οι πολίτε αυτοί το δικαίωμα, εφόσον δεν έχουν καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση, να μην καταγράφονται τα στοιχεία του. Γιατί να υπάρχει τέτοια μαζική εποπτεία και παρακολούθηση και τέτοιε πολιτικέ που να δικαιολογούν και να καλύπτουν του πάντε. Και όλο ιδιαιτέρω ε, η όθηση που δίνει το Συμβούλιο προ μια νέα πρόταση για την παρακολούθηση και την τήρηση δεδομένων σχετικά με τι επικοινωνίε, τι ε, ε, συνομιλίε των πολιτών, δεν είναι κάτι που αντίκειται στην διάθεσή μας και στην ελευθερία των μετακινήσεων για τα αρχαία των επιβατών. Κύριε Μπράιερ, καταλαβαίνω ότι είναι λεπτό το θέμα της στήριξης των δεδομένων. Είναι λεπτό και για την δική σας την ομάδα και αγγίζει και πολλές ευαισθησίες ε, εκτός της ομάδας σας. σε κάποιο βαθμό και σε περισσότερο από ότι σε κάποιο βαθμό μόνο, τη συμμερίζομαι. Ως πρώην ε, ευρωυπάλληλος ε, ανέκαθεν ε, τηρούσα την ομολογία και τις αποφάσεις, το περιεχόμενο δηλαδή, όσον έλεγε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι μας λέει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε ιδιαίτερα προσεκτικά. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε για να βρούμε λύσεις. Τώρα που γνωρίζουμε τι όρια έχει θέσει το δικαστήριο. Ε, πέραν αυτού, η δουλειά μας για την τήρηση των δεδομένων είναι κάτι που θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί από την πλευρά της Επιτροπής όταν έχουμε το σύνολο της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου στα χέρια μας, αλλά υπάρχουν και άλλες πολλαπλές δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκδίκασή τους. Έχω συζητήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ξέρω ότι θα αισθάνονταν μεγαλύτερη ασφάλεια εάν περιμέναμε την περάτωση και αυτών των υποθέσεων πριν ε, αποφασίσουμε τα περαιτέρω βήματα. Τώρα για τη γενικότερη ερώτησή σας. Το είπα δύο και τρεις φορές νομίζω ως τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκόσμιος πρωταθλητής για την προστασία των δεδομένων και του ιδιωτικού βίου. Είμαστε μια ομάδα στον κόσμο που έχουμε δώσει τις καλύτερες εγγυήσει στους πολίτες μας και ε, ισχύει μια αρχή που έχει οικουμενική αξία. Ε, η συγκατάθεση, η συνένεση του ανθρώπου, του ιδιώτη. Δεν πιστεύω ότι θα βαραβιάσουμε την αρχή αυτή σε κάποιες πτυχές των πολιτικών μας και σε κάποιες άλλες θα το δεχόμαστε είναι οικουμενική ισχύω αυτό. Είναι μέρο του ευρωπαϊκού τρόπου ζωή. Αυτό σημαίνει για μένα τουλάχιστον. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπρέιερ, έχετε δεύτερη ερώτηση. Σα ευχαριστώ για την απάντησή σα. Σεβασμό για τι αποφάσει του δικαστηρίου. Αυτό είναι ένα πράγμα. Όμω είναι κάτι διαφορετικό η λήψη πολιτικών αποφάσεων. Θέλετε να εφαρμόζετε τέτοιες ιδέες και σε υπο, ε, υποκείμενους τρόπους, σε υπόγειους τρόπους στήρισης και παρακράτησης των δεδομένων και μάλιστα με μαζική, ε, μαζικής εμβέλειας. Εδώ λοιπόν αυτό αφορά όλο τον πληθυσμό, το σύνολό του και στην απάντησή σας λέτε ότι το δικαίωμα για την ασφάλεια πρέπει να διαχωρίζεται από το δικαίωμα για την προστασία του ιδιωτικού βίου. Όμως αυτό δεν είναι σωστό, διότι δεν υπάρχει πουθενά το δικαίωμα ότι πρέπει κανείς να είναι ασφαλής από εγκληματική ενέργεια. Ε, Εσεί είστε και νομικό. Πώ μπορεί κανεί να μιλάει για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αν υπάρχει τέτοια παρανόηση στην ερμηνεία είναι πάρα πολλά τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου σας που δεν είναι εντελώς ε, ξεκάθαρα, όμως αυτό το δικαίωμα στην ασφάλεια πραγματικά μας προβληματίζει. Κύριε Σκηνά, ένα λεπτό για να απαντήσετε. Για το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να καθησυχάσει κανείς τους φόβους της ανησυχίας σας είναι εγώ και η Επίτροπος Γκάμπριελ μαζί, αλλά και η Επίτροπος Γιώχανσον, αν και νομίζω εγώ περισσότερο και από τους τρεις, ε, είναι να βεβαιωθούμε ότι όταν η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι πλέον έτοιμη από την Επίτροπο Βεστάγκερ και την, επίτροφο, την υποψήφια Επίτροπο Γκουλάρ, τότε σαφώς θα πρέπει να βρούμε τη σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ πολιτικής ε, ασφάλειας, υποστασίας και εγγύσεων. Δεν θεωρώ ότι πρέπει εδώ να υπάρξει ε, σχέση αντιφατική μεταξύ τους, σε αντιδιαστολή δηλαδή, ή κάποιο συντελεστή να έχει μηδενική τιμή για να κερδίζει κάποιο άλλο. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε στην πολιτική μα πρέπει να γίνει μέσω των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει ασφάλεια χωρί θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι εντελώ ξεκάθαρο. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν πρέπει να τα αντιληφθούμε όπω κάναμε ω τώρα, ω μια μελέτη αντικτύπου που πρέπει κάποια στιγμή να εκπαιδευτεί όπω το τέλο. Πρέπει να γίνει εγκαίρο στην αρχή, τη στιγμή που λαμβάνουμε την πολιτική απόφαση εξ αρχή. Ευχαριστώ. Και τώρα για τι επόμενε εξερωτήσει να δώσω το λόγο στον ε, συμπρόεδρό μου, τον ε, κύριο Λόπεθ Αγγιλάρ. Λοιπόν, ο συνάδελφο ε, Νίκολα Φέστ, ένα λεπτό παρακαλώ για την ερώτησή σα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Σχοινά. Στην αρχή είπατε ότι έχετε τρει στόχου Πρώτον, ε, προστασία της ισότητας ε, ανδρών και γυναικών, καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και τρίτον, η εφαρμογή του Παγκοσμίου Συμφώνου για τους ε, μετανάστες και τους πρόσφυγες. Αλλά υπάρχουν αντιφάσεις. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι ο Καρλ Λάγκερφελντ δεν ήταν ρατσιστής, ούτε λαϊκιστής, ούτε καν δεξιός. Αλλά με την κριτική που έκανε στην πολιτική της κυρίας ε, Μέρκελ που υποδέχθηκε τόσους πολύ, και είπε ότι δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε στη χώρα μας δύο εκατομμύρια μουσουλμάνους και παράλληλα να διαμαρτυρόμεθα για την άνοδο, την άνοδο του αντισημιτισμού. Πώς θα τα επιτύχουμε όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν από τη μία να θέλουμε να προστατεύσουμε την ισότητα ανδρών και γυναικών και τα δικαιώματα των και από την άλλη να υποδεχόμεθα τόσους ε, μουσουλμάνους. Από ποια μεριά λοιπόν είστε, μετανάστευση η προστασία των ε, ε, ομοφιλοφίλων Εβραίων και γυναικών. Δύο λεπτά κύριε Σχοινό. Ε, δεν ξέρω αν μπορώ να σας πω αυτά που σκέφτομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα προσπαθήσω. Φοβάμαι ότι έχετε δίκαιο. Κύριε Φέστ, με κάθε σεβασμό, δεν βλέπω ότι είναι είτε είτε. Απλά είναι διαφορετική άποψή μου. Καταλαβαίνω ότι ορισμένοι θέλουν, θέλουν να μας αναγκάσουν να σκεφτόμαστε έτσι. Εγώ δεν θα το κάνω. Εγώ θα αντισταθώ στον πειρασμό να σκεφτώ έτσι. Και πάω και λίγο μακρύτερα. Κοιτάζοντα προ αυτή τη μεριά. Επίση θα αντισταθώ στον πειρασμό αυτών που με πιέζουν Χρησιμοποιώντα αυτό το επιχείρημα να το κάνω. Αυτό ακριβώς θέλουν να επιτύχουν. Αυτή είναι ακριβώς η παγίδα που θέλουν να πέσουμε. Είτε, είτε. There are two There is... Δεν υπάρχουν δύο Ευρώπε. Υπάρχει μία Ευρώπη όπου ανήκουμε όλοι και υπάρχει χώρος για όλους. Αυτή είναι η απάντησή μου στον κύριο Φέστ. Άλλο ένα λεπτό κύριε Φέστ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σχοινά, βλέπω ότι ο Καρλ Λάγκεφελντ θα ήταν καλύτερος επίτροπος αντί για σας σε αυτή τη θέση. Και ελπίζω να είστε τόσο καλός μόδιστρος όπως αυτός. Ίσως να μπορέσετε να ακολουθήσετε μία στεναδρομία εκεί, γιατί εδώ δεν είστε κατάλληλος. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ κύριε Επιτροπέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσο χρόνο θέλετε. Αν θέλετε βέβαια. Όχι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Περνάμε στην επόμενη ε, ομιλήτρια, την κυρία Μελ Μπάρντε. Ένα λεπτό. Κύριε Σκηνά, ευχαριστώ πολύ για, την πολύ καλά διαρθρωμένη, για τις πολύ καλά διαρθρωμένες απαντήσεις σας και τις γραπτές και προ, τις προφορικές. Από την πολιστική πλευρά του χαρτοφυλακίου σας, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν μιλούμε για, τον, ένα, για ένα τρόπο ζωής ατόμων ή κοινοτήτων, ε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την έννοια της ταυτότητας. Έχετε κάποια πολιτική για την ταυτότητα και ποια θα μπορούσε να είναι αυτή. Πολύ σύντομοι ήσασταν. Συγχαρητήρια. Κύριε Σχοινά, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την ερώτηση για να απαντήσω και στην κυρία Ιντζήρ γιατί εκκρεμεί μια ερώτηση της. Α, έχει φυγεί από την αίθουσα, οπότε θα μείνω σε εσά μόνο. Όχι, δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη ταυτότητα. Προτιμώ να χρησιμοποιώ τη φράση κοινή αίσθηση του ανήκειν. Αυτή η έκφραση μας ε, καθησυχάζει όλους. Γιατί? Γιατί δίνει χώρο σε όλους. Εδώ είμαστε σε μια ήπειρο που όλοι έχουν πολεμήσει έναντι όλων των υπολείπων για κάθε δυνατό και πρακτικό λόγο. Ε, για ταυτότητες, για θρησκείες, ε, για εξαιτίας πολλώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τρομακτικό επίτευγμα και είναι επιτεύγμα γιατί καταφέραμε ε, να στηρίξουμε αυτό το οικοδόμημα σε ένα σύνολο αρχών, όπου όλοι, αν όχι όλοι οι περισσότεροι, νιώθουν άνετα. Το να ανοίξουμε την πόρτα της ε, πολιτικής ταυτότητας, των πολιτικών ταυτότητα δεν θα βελτιώσει απαραίτητα τις αυριανέ κοινωνίε. Οι αυριανέ κοινωνίε θα πρέπει να λειτουργούν χωρίς αποκλεισμού, να είναι ανθεκτικέ, να βασίζονται στις δεξιότητες, να έχουν πολιστικά εργαλεία και μια κοινή αίσθηση του ανήκειν. Δεν θα πρέπει να βασίζονται στο ότι εμείς είμαστε σε σύγκρουση ή αντίθετη με τους άλλους, όχι σε αντιδιαστολές. Αυτό θα ήθελα να αποφύγω. Η λέμε Μπάρντε για συμπληρωματική ερώτηση. Είτε χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ταυτότητα είτε όχι, υπάρχει μία λέξη κλειδί που λείπει από τις απαντήσεις σας και από τις αρμοδιότητές σας. Είναι η έννοια της ευρωπαϊκής ιστορίας και η κοινωνική μνήμη. Στην τελευταία του σύνοδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, υιοθέτησε ένα ψήφισμα για την, ε, τη μνήμη, την ευρωπαϊκή μνήμη για ένα καλύτερο μέλλον. Ε, πώς θα το εφαρμόσετε αυτό το ψήφισμα. Ένα ακόμα λεπτό στον κύριο Σχοινά. Δεν θα έπρεπε να απευθύνεται αυτή την ερώτηση σε μένα. Δεν χρειάζεται εγώ να αναλάβω αυτή την ευθύνη της, ευθύ, της ιστορίας της δημοκρατίας των αρχών. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα της κυρίας Σουίτσα, που νομίζω βρίσκεται σε μια διπλανή αίθουσα αυτή τη στιγμή και έχει στο και ό,τι τα θέματα της δημοκρατίας και της δημογραφίας, καθώς επίσης και στις αρμοδιότητες της κυρίας Γιούροβα, που έχει την ευθύνη των θεμάτων σχετίζονται με τις αρχές και την οποία θα ακούσετε την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε καλό είναι να μην μπω στο δικό τους γήπεδο. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Λισάβετ Βόσεμπερκ Μπριονίδη. Καλησπέρα κύριε Σχοινά, σας εύχομαι καλή επιτυχία θα αναφερθώ στην συμφωνία δήλωση ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας που εδώ και τέσσερα χρόνια λειτουργήσε σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικά μειώθηκαν σημαντικά οι ροές και μπορέσαμε να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων στη μεσόγειο. παρά τα τελευταία υπάρχει μια δραματική αλλαγή των πραγματικών περιστατικών. Οι δεκάδες άνθρωποι έρχονται από τα παράλια της Τουρκίας. Η αύξηση των ροών είναι της τάξης του 200% από το Μάιο μέχρι σήμερα και αντιλαμβάνεστε ότι για τη χώρα μας την Ελλάδα, που είναι χώρα πρώτης υποδοχής, η κατάσταση είναι δραματική και μη διαχειρίσιμη η Τουρκία είχε αναλάβει την υποχρέωση στη συμφωνία αυτή να αποτρέψει το άνοιγμα καινούριων οδών, καινούριων δρόμων και στη θάλασσα και στην ξηρά και να συνεργαστεί τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με τις τρίτες χώρες. Φαίνεται ότι αυτό στην πράξη έχει προβλήματα πώς αξιολογείτε την λειτουργία της δήλωσης συμφωνίας μέχρι σήμερα και αν πιστεύετε ότι πρέπει να ασκηθούν πιέσεις προς την Τουρκία να ε, υποχρεωθεί να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Your time to respond, two minutes. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά για την απάντησή σας. Κυρία Βόζεμπερκ, νομίζω ότι η, η αφετηρία ε, της απάντησης σε αυτό το θέμα πρέπει να είναι η παραδοχή εκ μέρους μας ότι η Τουρκία φιλοξενεί εδώ και χρόνια στο έδαφος της πάνω από 3 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες. Είναι ένα βάρος που έχει αναλάβει και για το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί. Όπως πρέπει να αναγνωριστεί και ο Λίβανος και η Ορδανία, κράτη που έχουν αναλάβει δυσανάλογα μεγάλα βάρη και τιμούν τις υποχρεώσεις τους προς τους ε, αδύναμους και τους ζητούντες άσυλο. Είναι αλήθεια ότι η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας παρήγαγε μέχρι πρόσφατα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ουσιαστικά ε, εκμυδένισε τις ροές σε ένα ποσοστό μεταξύ 85% και 90%. Είναι επίσης γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ γενναιόδωρα με ένα ποσό που ε, φτάνει τα 6 δισεκατομμύρια σε δύο προγράμματα έχει αναλάβει ουσιαστικά τη χρηματοδότηση του βάρους υποδοχής αυτών των απελπισμένων ανθρώπων που βρίσκονται στην Τουρκία. Είναι επίσης αλήθεια ότι μερικές πλευρές της συμφωνίας έμειναν εκρεμείς. Αυτά είναι τα δεδομένα. Όπως είναι επίσης αλήθεια ότι η τελευταία επιθετική ρητορική που συνδέεται με τις εξελίξεις στη Συρία και στον Ιτλίμπ επιβαρύνει την κατάσταση. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναεπισκεφθούμε τη συμφωνία, να την ξαναφρεσκάρουμε. Είναι πολύ θετικό ότι as we speak που λένε, τη στιγμή που βρισκόμαστε ο Επίτροπος Αβραμόπουλος μαζί με τον Υπουργό Ζήχοφα και τον Υπουργό Καστανέ βρίσκονται στην Τουρκία ακριβώς για αυτό το θέμα και αύριο θα πάνε στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό να αναλάβει η Τουρκία να καταλάβει το ρόλο που έχει ως εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση αυτού του προβλήματος που είναι κοινό και για τους δυο μας και είναι σημαντικό και η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές αρχές να αναλάβουν ότι κάποια από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε ελληνικό έδαφος για την καλύτερη διαχείριση των αρνητικών συνοπιών, δηλαδή τις μη γρήγορε επιστροφές, μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί όπως ξέρετε, πιστεύω μέσα από αυτή τη λογική θα βρούμε μια άκρη στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Back to you, Mrs. Εσεί πάλι, κυρία Βόζεμπεργκ, για τι συμπληρωματική σα ερώτηση. Ε, κύριε Σκινά, σα ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και τι διαπιστώσει σα συμφωνώ. Όπω φαντάζομαι και εσεί συμφωνείτε, ότι η αλλαγή είναι δραματική του τελευταίου μήνε. Ε, υπάρχει ένα καινούριο δεδομένο, υπάρχει μια καινούρια κυβέρνηση στη χώρα μα που έχει μια διαφορετική μεταναστευτική πολιτική, η οποία εναρμονίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη συμφωνία. Με το δεδομένο που είπατε ότι θα ξαναδούμε τη συμφωνία, Θέλω να σας ρωτήσω, θα τη δούμε από μηδενική βάση ή εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, κάποιες βελτιώσεις που να δεσμεύουν και τα δύο μέρη να τηρούν τις υποσχέσεις τους και τους όρους της συμφωνίας αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε τον λόγο, κύριε αλλά νομίζω ότι η απάντηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επίσκεψη Αβραμόπουλου Ζιχόφερ στην Άγκυρα σήμερα το βράδυ. Ε, μόλις ε, θυμήθηκα ότι ο Υπουργός ε, Καστανέρ νομίζω δεν ταξίδεψε λόγω της, ε, ε, της επίθεσης στο Παρίσι. Ε, όντως πρέπει να δούμε με την τουρκική κυβέρνηση τι ακριβώς μπορεί να αποτελέσει το κέντρο αυτής της φρέσκιας οπτικής στη δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκίας. Δεν θέλω τώρα να προτρέξω. Νομίζω μιας και το θέτετε ότι είναι η ώρα να πούμε ότι η Ελλάδα δεν θα αφαιθεί μόνη της στη διαχείριση αυτών των ροών. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αφαιθεί μόνη της. Είναι ευχή έργο αυτή τη στιγμή που η, ελληνική κυβέρνηση, η νέα ελληνική κυβέρνηση ευθυγραμμίζει σε μεγάλο βαθμό τις ε, δράσεις της με τις ευρωπαϊκές πολιτικές μετανάστευσης και ελπίζω ότι από αύριο, σε αυτές τις λίγες που μας μένουν, θα μπορέσουμε να δρομολογήσουμε αυτή τη νέα ματιά στην Ευρωτουρκική Συμφωνία θετικά που θα ξεπερνάει ρητορικέ και λόγια και απειλέ. Νομίζω ότι αυτά πια δεν έχουν καμιά σημασία στη διαχείριση του θέματος που μας απασχολεί. Thank you Και πάλι σας ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Κελέρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε. Η θανατηφόρα πυρκαγιά στο, στο καταβλισμό της Μόριας, στη Λέσβο, την περασμένη Κυριακή, μας θυμίζει ότι πρέπει η Ευρώπη κατεπηγόντως να προβλέψει ένα κοινό σύστημα ασύλου. Μιλήσατε για ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Μια συνένεση, μια συμφωνία για μια νέα αρχή Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα κύριε Σχοινά, μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβετε, ιδίως για το πακέτο του ασύλου. Τι ηθής, τι η χαρακτήρα θα, έχει, θα είναι αυτό το πακέτο, ποια εργαλεία προβλέπετε και τι χρονοδιάγραμμα διαβλέπετε. Ευχαριστούμε κύριε Σχοινά. Ευχαριστώ κυρία Κελέρ για την ερώτησή σα, Θα προσπαθήσω να σας πω όσο περισσότερα μπορώ δεδομένου ότι όπως συμφωνήσαμε με την Ήλβα Γιώκανσον πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε και κάποιες συνεννοήσεις, να πάμε και σε όλες τις πρωτεύουσες για να συζητήσουμε, να αφουγκραστούμε τις δικές σας απόψεις, να έχουμε μια σφαιρική εικόνα και μετά να κάνουμε συγκεκριμένε προτάσεις. Τώρα δεν θέλουμε να αποτύχουμε. Δεν πρέπει να αποτύχουμε. Μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή, είναι μια ευκαιρία, αλλά τώρα failure is not an option. Δεν υπάρχει ε, ε, περιθώριο για αποτυχία. Πρέπει να πετύχουμε. Θα προσπαθήσω λοιπόν εντό αυτών των ορίων που σας έθεσα να σας πω εγώ προσωπικώς τι πιστεύω για τη βάση αυτής, αυτού του συμφώνου. Το είπα και στην κυρία Μιτσόλα στην αρχή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διατηρήσουμε τα πέντε νομοθετικά κείμενα και τα βήματα πρόοδου που αυτά μας επέτρεψαν να επιτελέσουμε. Αυτό για μένα είναι το σημείο αφετηρίας. Αυτά παραμένουν ω βάση. Δεύτερον, πρέπει να επικεντρωθούμε στα δύο κείμενα που λείπουν, Δουβλίνο και διαδικασίες. Ε, η μεταρρύθμιση του Δουβλίνου και οι διαδικασίες. Γιατί, Γιατί το σύστημα ασύλου μας ε, ε, έχει ως, βασίζεται στη λογική μιας διαφορετικής Ευρώπης. Δηλαδή, ε, ασύλο για κάποιους που ξέφευγαν από την δικατορία στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία. Τώρα έχουμε ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα διαφορετικών διαστάσεων. Δεν μπορούμε να ζούμε με το παλιό σύστημα ασύλου στη σημερινή εποχή. Αλλά για να απεγκλωβιστεί η κατάσταση, η διάθεση από τα κάτι μέλη που μπλοκάρουν το κείμενο και να κάνουμε μια νέα αρχή πρέπει να συγκεντρώσουμε και κάποιες άλλες παραμέτρους. Πρέπει να υπάρξει η επιστροφή και οι διευθετήσεις, οι συμφωνίες για την επανεισδοχή είναι θεμελιώδου σημασία. Πρέπει να ξαναδούμε τον κανονισμό Σέγγεν. Διότι η εσωτερική ελευθερία, η ελευθερία τη κυκλοφορία, ε, έχει να κάνει και με το πώ προστατεύουμε τα σύνορά μα. Πρέπει να ξαναδούμε λοιπόν τη διάσταση των σύνορων και την νόμιμη μετανάστευση. Πιστεύω ότι με όλα αυτά τα στοιχεία μπορούμε να έχουμε όσα οπωσδήποτε χρειαζόμαστε για μια νέα αρχή. Κυρία Κελέρ, και πάλι ένα λεπτό. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, ευχαριστώ. Το είπατε. Καθυστερεί πάρα πολύ η μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου. Θυμόμαστε το 2016 ήδη υπήρχαν νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν επέτρεψαν να καταπραίνουν τις εντάσεις και τις διαφωνίες μεταξύ κρατών μελών. Θυμάστε στο Κοινοβούλιο η προηγούμενη θητεία εργάστηκε σκληρά για να πετύχει μια ευρία πλειοψηφία. Η ερώτησή μου λοιπόν και επιμένω το χρονοδιάγραμμα. Πώς προτίθεστε να προχωρήσετε για το θέμα αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η αναποφασιστικότητα ή μάλλον η απουσία απόφασης ουσιαστικά επιτρέπει να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες. Δεν προχωρούμε. Λόγου χάρη θα παροτρύνεται το Συμβούλιο να εφαρμόσει τους κανόνες της ενισχυμένης πλειοψηφίας που μπορούν, ε, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε αυτόν τον χώρο. Κύριε Σκινά, ένα λεπτό για να συμπληρώσετε την απάντησή σας. Μια εύκολη απάντηση και μια κάπως δυσκολότερη. Η εύκολη απάντηση είναι για το χρονοδιάγραμμα. Η πρόθεσή μας, σε συνεργασία με την αρμόδια υποψήφια επίτροπο, είναι μετά από αυτήν την ε, συνεννόηση με τι πρωτεύουσε πολύ γρήγορα μέχρι το τέλο τη χρονιά να μπορούμε να σα υποβάλουμε, όπω λέμε στα γαλλικά, ένα ε, scoping paper, ένα uh, έγγραφο, ένα σημείωμα που να καλύπτει τι βασικέ πτυχέ, uh, βολιδοσκόπηση α πούμε. Και μετά, αφού γίνει αυτό και αν όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι με τον ενθουσιασμό όλου του κολεγίου και τη συμμετοχή όλων και της ε, Προέδρου θα ξεκινήσουμε στην αρχή της επόμενης χρονιάς. Ναι, μπορείτε, μπορείτε, έχετε ακόμη χρόνο. Για τη δύσκολη απάντηση τώρα. Λέτε, πρέπει να ανατρέξουμε στην ενισχυμένη πλειοψηφία. Κέρια σημασίας η ερώτηση, αλλά δύσκολη η απάντησή της. Γιατί, Γιατί προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ενισχυμένη ε, πλειοψηφία με την επιτόπου ε, εγκατάσταση και τους σχετικούς κανόνες. Ίσως τότε καταφέραμε να λύσουμε το πρόβλημα εν μέρη, όμως η ενισχυμένη πλειοψηφία άφησε τραύματα ε, και πληγές δημιούργησε δυστυχώς ε, πληγές της επούλωτες. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε μια νέα αρχή. Ναι, από τεχνικής πλευράς αυστηρός θεωρητικά υπάρχει ενισχυμένη πλειοψηφία. Αλλά από πολιτικής σκοπιάς είναι προτιμότερο να την αποφύγουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ένα λεπτό ο κύριος Κώστας Παπαδάκης. Παρακαλώ. Κύριε Σχοινά, η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσφυγικό μεταναστευτικό χαρακτηρίζεται από την αντιδραστική κατεύθυνση των απελάσεων, που έβυχα αποκαλείται επιστροφέ, τη ενίσχυση των στρατιωτικών μέσων στα σύνορα, τη μετατροπή σε κανόνα τη κράτηση για ανθρώπου που εξαναγκάστηκαν κάτω από συνθήκε πολέμου, υπερελιστικών επεμβάσεων και εξαθλίωση να εγκαταλείψουν την πατρίδα του, και είναι δε ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη ο επιχειρούμενος περιορισμός και η ίδια η αλλίωση της έννοια του πρόσφυγα. Στην Ελλάδα η νέα κυβέρνηση σε συνέχεια της προηγούμενης προωθώντας την ίδια ευρωενωσιακή κατεύθυνση προεξοφλεί κιόλα με ανακοινωθέντα στόχο 10.000 απελάσεις ως το 2020. Επίσης, μεταξύ άλλων, να πάψουν οι πρόσφυγες με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής να συμπεριλαμβάνονται στις ευάλωτες ομάδες ετούντων άσυλο. Οι παραπάνω ευθείες παραβιάζει διεθνών αναγνωρισμένων δικαιωμάτων συνιστούν την αποκαλούμενη προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής ή και πολύ χειρότερα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηματοδοτείται μέσα από αυτά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Σκηνά. Κύριε Παπαδάκη, ε, μου δίνει την ευκαιρία να επαναλάβω κάτι που είπα στην αρχή. Ε, σέβομαι όλες τις απόψεις και όλες τις προτάσεις που έχουν μια τάση να ερμηνεύουν το πολύ σύνθετο μεταναστευτικό ε, φαινόμενο από μια συγκεκριμένη οπτική. Ειλικρινά σας λέω ότι σέβομαι και πιστεύω ότι έχουν και μια παραγωγική συνεισφορά στο, στο θέμα. Αλλά δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση. Η Ευρώπη βρίσκεται στο κέντρο αυτού του μεταναστευτικού φαινομένου που μας ε, είναι απαραίτητο να σκεφτούμε συνολικά. Πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Και αυτά που θέλουμε και αυτά που ενδεχομένως δεν θέλουμε. Τώρα, αν σας καταλαβαίνω καλά, μου λέτε ότι ε, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, κάνοντας δηλαδή και άσυλο και επιστροφές και διαχείριση ροών, ε, κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι εναντίον των ε, αξιών μας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Θα ήταν εναντίον των αξιών μας αν η Ευρώπη ακολουθούσε το μοντέλο της Αυστραλίας. Αυτοί που θέλουν τον Αυστραλιανό τρόπο ζωής θα θέλουν και το Αυστραλιανό μοντέλο διαχείρισης της μετανάστευσης. Δεν είναι ο δικός μας τρόπος. Εμείς κάνουμε τα πράγματα αλλιώς. Τα κάνουμε συνολικά, με όλες τις παραμέτρους που έχουμε στα χέρια μας. Είμαστε κοινωνίες και κράτη-μέλη δικαίου. Όλα μας τα κράτη-μέλη σέβονται τις διεθνείς συνθήκες τις Γενέβης, όλα μας τα κράτη-μέλη σέβονται τη διεθνή και ευρωπαϊκή ένωμη τάξη. Δεν βλέπω δηλαδή, με συγχωρείτε κιόλα, δεν βλέπω γιατί πρέπει αυτό αμέσως να μεταφραστεί ότι τα πράγματα είναι στραβά. Εγώ δεν τα βλέπω στραβά. Δεν τα βλέπω όλα λιμένα, αλλά βλέπω μια συνεπή ευρωπαϊκή προσπάθεια να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε σύμφωνα με τις δικές μας αξίες. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδάκη, παρακαλώ ένα λεπτό για συμπληρωματική. Κύριε Σκινά, δεν ισχυρίστηκα ότι αυτά που περιέγραψα είναι ενάντια στι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ είναι οι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ευρωπαϊκό τρόπο ζωή είναι η μόρια, είναι τα hot spot. Και με δεδομένο ότι εδώ και 3,5 χρόνια η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι επιβάλλει το μαζικό εγκλωβισμό προσφύγων στα ελληνικά νησιά, αυτέ τι μέρε στην Ελλάδα κλείσεται μια δραματική και συνάμα εκρηκτική κατάσταση και ε, επί της ουσίας δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες ζουν σε άθλιες συνθήκες, όχι μόνο στη Μόρια αλλά και στα άλλα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας, οξύνοντας τα προβλήματα και για τους ντόπιου κατοίκους. Πώς λοιπόν τοποθετήσετε στο γεγονός ότι πλέον αποδεικνύεται ότι ο ισχυρισμός μέχρι τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της πως η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σταματούσε τις ροές έχει στην πράξη καταρρεύσει. Πώ επίση τοποθετήσετε στην ανάγκη να κλείσουν εδώ και τώρα όλα τα hot spot και να υπάρξει μεταφορά των προσφύγων και μεταναστών στην υπηρετική Ελλάδα σε αξιοπρεπεί και δημόσιε δομέ φιλοξενία με προοπτική τη γρήγορη μεταφορά του στι χώρε πραγματικού προορισμού του με πλήρη τήρηση των δικαιωμάτων για το άσυλο. Σα ευχαριστώ. Thank you. Now your minute to close. Παρακαλώ, ένα λεπτό για να ε, ολοκληρώσετε την απάντησή σας στην ερώτηση αυτή, κύριε Σκηνά. Είναι λίγο το ένα λεπτό για όλα αυτά τα θέματα που έθεσε ο κύριος Παπαδάκης, αλλά ίσως πολύ γρήγορα πρέπει να πω ε, ε, μερικές από τις επιτυχίες μας, κύριε Παπαδάκη, που νομίζω ότι τις ε, υποτιμήσατε. Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι οι 700.000 ψυχές που σώθηκαν στη Μεσόγειο, χάρη σε εμά. Είναι οι γιαγιάδες της Λέσβου, είναι η επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα και στη Λέσβο που χαιρετίζει τις ευρωπαϊκές αξίες. Είναι όλα έσω έχουμε κάνει στο άσυλο, ότι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, ξέρετε ότι το 2015 και 2016 δεν υπήρχε τίποτα στα νησιά του Αιγαίου και ξεκινήσαμε από το μηδέν. Τώρα αν με ρωτήσετε ότι η κατάσταση στη Μόρια με ικανοποιεί, εγώ είμαι ο πρώτος που σας πω ότι δεν με ικανοποιεί. Με πληγώνει και ως Έλληνα και ως Ευρωπαίο. Αλλά δεν πέφτω στην παγίδα να εκτιμήσω ότι είναι αποτέλεσμα μιας παραμέτρου αυτό. Αυτό είναι ένας πολυπαραγοντικός, μια πολυπαραγοντική εξίσωση, στην οποία πρέπει να σκεφτούμε πώς στάσαμε τα τελευταία τρία χρόνια. Το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θα το δούμε και η Ευρώπη, όπως είπα πριν, θα είναι ε, αρρωγός στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Τώρα ένα λεπτό ο Στάλφος Λούκατς Τσκόκου. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Σχοινά, θα συντονίσετε την εργασία μιας, ενός φιλοδόξου θεματολογίου για την εκπαίδευση. Πώς θα βοηθήσετε την εκπαίδευση των ενηλίκων μέσω του νέου στρατηγικού πλαίσιου. Και δεύτερον, πώς θα διασφαλίσετε ότι οι άτυπες μορφές ε, μάθησης για τους ε, ε, ενηλίκους, για τους ενήλικες θα προωθηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά κύριε Σχοινά. Ευχαριστώ κύριε Κόκο. Πολύ σημαντική ερώτηση. Συμπληρώνει τα θέματα που έθιξαν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Απασχόλησης. Κοιτάξτε, πρέπει να συνδέουμε τις δεξιότητες με την αγορά εργασίας και μέσω ήπιων δεξιοτήτων να βοηθάμε την ένταξη των ευαλώτων κοινωνιών και να βελτιώνουμε τις δεξιότητες. Αλλά τώρα θέτω το θέμα της διαβίου κατάρτισης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Θα έλεγα ότι είναι μία από τι κύριε προτεραιότητε μα. Γιατί η περίοδο όπου οι Ευρωπαίοι εκπαιδεύονταν ως νέοι και μετά δεν χρειάζονταν, δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο, έχει περάσει. Η δική μου γενιά εκπαιδεύτηκε μόνο σε ένα πράγμα ως τελευταία γενιά για να συνοδεύσουμε τη διαβίου κατάρτιση πρέπει να έχουμε ένα συνολικό ε, οπλοστάσιο και ήδη έχουμε σημαντικά εργαλεία στη διάθεσή μας. Για παράδειγμα η κυρία Γκάμπριελ στις αρμοδιότητές της. Για παράδειγμα το έρασμο συν και αυτά που περιέχει αλλά και αυτά που περιέχει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να εντοπίσουν τις ανάγκες τους στο θέμα της διαβίου κατάρτισης. Γιατί μια άλλη τάση είναι η εξής. Εκπονούμε προγράμματα εμείς στις Βρυξέλλες με τρόπο, πώς να πω, με μια οργανωτίστικη λογική, δηλαδή προγράμματα που είναι ίσο, εύκολα να τα διαχειριστούμε, να τα πληρώσουμε, και μετά διαπιστώνουμε ότι δεν είναι τα κατάλληλα για τις ανάγκες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Τονίζω ότι πρέπει να έχουμε μια αντίστροφη προσέγγιση. Από κάτω προ τα πάνω. Πάμε στα κράτη-μέλη να εντοπίσουμε τι ανάγκε και κατόπιν να τα αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι ανάγκε μέσω, μέσω πολιτική. Κύριε Κόχουτ, παρακαλώ, για να συμπληρώσω την ερώτησή σα. Παρακαλώ. Είπατε ότι θέλετε να υπάρχει περισσότερη πρόσβαση για όλα τα τμήματα της κοινωνίας στην κατάρτιση και ιδιαίτερα για τις μειονότητες και τα άτομα με αναπηρίες. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτό. Πώς θα ενθαρρύνετε τις κυβερνήσεις να σας βοηθήσουν. Για παράδειγμα την ε, πολωνική και ουγγρική κυβέρνηση. Πώς θα τις ενθαρρύνετε να τα κάνουν αυτά. Έχετε δίκιο όπως εντοπίζετε τα προβλήματα. Δεν θα είναι εύκολο, συμφωνώ. Όπως ξέρετε, για να μην υπάρχουν διακρίσεις, κυρίως χρειάζεται ομοφωνία. Ούτε αυτό βοηθάει. Έχουμε την οδηγία, την οριζόντια αυτή οδηγία κατά των διακρίσεων και είμαι περήφανος που ως Ευρωβουλευτής το 2008 την υπερψήφισα παρά το ότι το κόμμα μου ήταν κατά. Ρομπέρτα με συγχωρείς, ε, απειθάρχησα ως προς την ε, κομματική γραμμή τότε. Αλλά είμαι περήφανο που ψήφισα υπέρ αυτή τη οδηγία, η οποία έκτοτε έχει κολλήσει στο Συμβούλιο. Άρα σωστά εντοπίστε το πρόβλημα. Αλλά χαίρομαι που η Φιλανδική Προεδρία τώρα κάνει μια τελική προσπάθεια για να ξεπεράσει το αδιέξοδο. Ξέρω ότι στις, 28, ε, στις 24 Οκτωβρίου υπάρχει ένα Συμβούλιο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Εάν η Φιλανδική Προεδρία καταφέρει να ξεπεραστεί το αδιέξοδο για αυτό το θέμα, τότε θα είναι μια πρώτη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναδίνω την Προεδρία στην συνάδελφό μου της Επιτροπής Πολιτισμού. Για τις τελευταίες ερωτήσεις ε, έχουμε καταρχήν τον Γερούν Λενάρς του ΕΛΚ από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο αριθμός των αμφίξεων έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κοντά στο να αντιμετωπίσει μια μελλοντική κρίση. Το έχετε πει και στο παρελθόν, το είπατε και σήμερα, η μόνη πραγματικά καλή προσέγγιση στη μετανάστευση είναι η ολιστική ε, καλές πολιτικές ασύλου, διαδικασίες, ε, έλεγχος των συνόρων, συνεργασία με τρίτες χώρες κλπ. Αλλά λείπουν οι επιστροφές. Μόνο το 1 τρίτο των ατόμων τα οποία δεν έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας ε, επιστρέφουν. Αυτό σημαίνει ότι τα 2 τρίτα αγνοούν τις διαδικασίες μας και παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρανόμως. Αυτό πλήττει και την στήριξη που χρειαζόμαστε από την κοινωνία. Οι επιστροφέ μπορούν να γίνουν μόνο αν συνεργαστούμε με τρίτες χώρε. Δυστυχώ αυτό είναι και το κομμάτι τη πολιτική στο οποίο δεν έχουμε να δείξουμε πολλέ επιτυχίε στο παρελθόν. Οπότε η ερώτηση είναι πώ πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία με τρίτες χώρε και ποια συγκεκριμένα βήματα σκοπεύετε να λάβετε προ αυτήν την κατεύθυνση. Ο λόγος του κύριο Σχοινά για δύο λεπτά. Κύριε Λενάρης, πραγματικά αγγίζεται ένα από τα καινούρια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να φέρουμε στο σύμφωνο ε, ασύλου και μετανάστευσης. Να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για μια καινούρια αρχή. Στην ε, ε, επιστολή καθηκόντων μου είναι ότι μία από τις προτεραιότητές μου θα είναι μαζί με την ε, Γιωτόρ Πιλάινεν που είναι η υπεύθυνη για τις ε, διεθνείς εταιρικέ σχέσεις να ξεκινήσουμε στην αρχή της θητείας μας ήδη ένα καινούριο κύμα συμφωνιών επανεισδοχής και διευθετήσεις με χώρες προέλευσης και χώρες διέλευσης. Το χρειαζόμαστε. Ε, δεν μπορούμε να προσποιούμε θα ούτε συμβαίνει. Ε, οι επιστροφές έχουν σχέση με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αλλά πέραν αυτού χρειαζόμαστε καινούριε εταιρικέ σχέσεις με αυτές τις χώρες, ε, προς όφελος και των δύο πλευρών. Θα ήταν λάθος να χτίσουμε αυτές τις συμφωνίες επανεισδοχής μόνο βασισμένη σε μια σε ένα τμήμα της πραγματικότητας που έχει σχέση με μετανάστευση. Έχουμε πολλά κοινά και έχουμε πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να τις βοηθήσουμε αυτές τις χώρε. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα έξυπνα και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Οι συμφωνίες επανεισδοχής θα πρέπει να έχουν νόημα και για τις τέτοιε χώρε και για μα, αλλά όχι μόνο για μα. Και έχουμε αρκετά εργαλεία, θεωρήσεις, ήπια ισχύ, χρήματα, υποτροφίες, εμπόριο, εκπαιδευτική συνεργασία. Όλα αυτά μπορούν να μπουν στο τραπέζι στη διαπραγμάτευση αυτών των συμφωνιών επανεισδοχής. Χωρίς τέτοιες συμφωνίες μην περιμένετε βελτίωση κύριε Λέναρης. Αυτά πάνε μαζί και θα αποτελέσουν τμήμα του νέου συμφώνου. Thank you very much. Ε, κύριε Λέναρς, συμπληρωματική ερώτηση. Συμφωνώ στα όσα είπατε για τις επανεισδοχές και πολύ καλό να ξεκινήσουμε με ένα περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων χωρών στόχων. Και τα επόμενα πέντε χρόνια θα σας βοηθήσει πολύ και είπατε εκπρόσωπος καθώς επίσης και Υπουργή Εξωτερικών των κρατών μελών Μόνο έτσι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί από τα τελευταία πέντε χρόνια. Ελπίζω να την έχετε. Τώρα, οι αμοιβώ ωφέλιμε εταιρικέ ε, ε, συμφωνίες ε, δεν είναι ευθυνέ και δεν το λέω αυτό μόνο επειδή παντρεύτηκα πρόσφατα. Τι θα γίνει με το Ταμείο Ασύλου μετανάστευση και ενσωμάτωση, το ΑΜΙΦ, πώ θα χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να σα βοηθήσει να συνάψετε τέτοιου είδου συμφωνίε με τρίτε χώρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Χινά για ένα λεπτό. Θα είμαι σύντομος, ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο Γέρον. Έχεις δίκιο. Που λες ότι ναι, πρέπει να ξεκινήσουμε με καινούριο ενθουσιασμό και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε με αυτά τα εργαλεία που διαθέτουμε. Τόσο ό,τι αφορά τα κονδύλια και τους πόρους. Ε, οι πόροι δεν είναι μόνο χρήματα, την άλλη μεριά έχουμε και άλλα πράγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, ω μοχλούς στις συζητήσει μας με αυτές τις τρίτες χώρες. Είπα, Θεωρήσει εμπόριο, συνεργασία, επενδύσεις, εκπαίδευση. Τώρα, από την πλευρά των κονδυλίων. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε αυτό το καινούριο πρόγραμμα που δεν μπορώ καν να το προσφέρω, NCCI, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τώρα πώς ούτε καν πώς λέγεται. Ε, αυτό θα μας ε, δώσει αρκετά χρήματα ώστε να αντιμετωπίσουμε και τις αιτίε και τις πραγματικές αναπτυξιακές ε, ανάγκες ε, και τα πόσα που χρειαζόμαστε για την εγγύηση των ασφάλιση των συνόρων. Σα ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο στον καταλογό μα των αγορητών, ο κύριο Κιζιλ Γιούρεκ από την Επιτροπή Πολιτισμού. Κύριε Σχοινά, σε ε, διαστολή με όσα αναφέρει το χαρτοφυλάκιό σα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα τρόπο ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμω πολιτικέ αρχέ για την προστασία τη αξιοπρέπεια, τη πολυφωνία, τη επικοινομορφία, τη ισότητα, τη δικαιοσύνη και ε, ζούμε σε μια περίοδο όντω όπου ε, εντείνεται ο φιλετικό ρατσισμό. Τι θα, μέτρα θα λάβετε για να αντιμετωπίσετε τι προκλήσει που προκύπτουν λόγω του πολιτιστικού αυτού ε, ρατσισμού, στι γραπτέ σα απαντήσει, κυρίε λέτε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, και παραθέτω εδώ το κείμενο, ε, είναι ε, ριζωμένο στην κουλτούρα μας και στον πολιτισμό μας και πρέπει να τον προστατεύσουμε. Εδώ λοιπόν για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό λέτε ότι πρέπει να προστατεύσουμε το αγαθό αυτό. Από ποιον, από ποιον πρέπει να πιστέψουμε τον ευρωπαϊκό, να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τον θεωρείτε ανώτερο. Και λέτε ότι δεν σας αρέσουν οι ισμοί και ο φεμινισμός ε, είναι, ε, ο φεμινισμός είναι μια, ένας σεισμός. Δεν σας αρέσει ούτε αυτός ας πούμε. Ξεκινώ με τον φεμινισμό. Πιστεύω στην ισότητα των φύλων. Είναι το ίδιο και δεν μιλάμε και με ισμό. Κύριε Κιζιλγιουρέκ, να συνεχίσουμε με την ερώτησή σας. Δεν είμαι βέβαιος τι εννοείται με τον πολιτιστικό ρατσισμό. Πώς το αντιλαμβάνεστε. Προσπαθώ να καταλάβω ότι θα δικαιολογούσα τη χρήση ενός τέτοιου όρου σε αυτό το κοινοβούλιο. Πού είναι ο πολιτιστικός ρατσισμός. Ε, μεταφραζόμαστε σε 23 γλώσσες ταυτόχρονα. Έχουμε συμμετέχοντες εδώ ανθρώπους από όλες τις προελεύσεις. Γλωσσικές, θρησκευτικέ, φιλετικές που έχουν εκλεγεί απευθείας από τον κόσμο της Ευρώπης. Πού είναι ο πολιτιστικός ρατσισμός. Εγώ βλέπω πολιτιστικό πλούτο και βλέπω και πολιτιστική υπερηφάνεια όταν ακούω ανθρώπους σαν εσάς, σαν την κυρία Ισμικ, τον ε, κύριο Μάτζιντ, πού είναι ο πολιτιστικός ρατσισμός. Δεν έχω γνωρίσει εγώ αυτή την ε, έννοια, ούτε καταλαβαίνω και τι είναι. Όταν κοιτάζω τα εργαλεία μας, όταν βλέπω τα προγραμματά μας, το, τη Δημιουργική Ευρώπη, το Creative Europe, το Erasmus και ούτω καθεξής, βλέπω ότι έχουμε το αντίθετο από αυτό για το οποίο μας κατηγορείτε. Ότι φέρνουμε τον κόσμο πέρα από τα σύνορα για να πάρουν αυτό που θέλουν. Ταξίδια, σπουδές, ε, απασχόληση, εμπόριο. Πού είναι αυτός ο πολιτισμός του ρατσισμού στην Ευρώπη. Πραγματικά θα ήμουν πολύ περίεργος να πάω και να το δω κάπου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει φόβος ε, κάποιας, ε, κάποιου δεσπόζοντος πολιτισμού, κάποιου πολιτισμού που να υπερτερεί, κάποιου που να είναι πρώτος. Αλλά νομίζω ότι η δύναμή μας, όπως σωστά είπατε στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ε, η δύναμή μας είναι η ποικιλομορφία στις αξίες, στις γλώσσες μας, τον τρόπο που ζούμε. Όταν λοιπόν λέω ευρωπαϊκός πολιτισμός και λέω ότι τον ζηλεύουν στον υπόλοιπο κόσμο, Λέω ότι όταν είναι κανείς στην Κίνα θέλει να πάει στο Λούβρο, θέλει να πάει στον Παρθενώνα, θέλει να επισκεφθεί την πολιτιστική μα κληρονομιά. Αυτό εννοώ. Μας ζηλεύουν, μας εποφθαλμιούν, δεν εννοώ αποκλεισμό, δεν εννοώ εμείς ε, κατά εναντίον των άλλων. Με παραμηνέυσατε και με παρανοήσατε πολύ βαθιά αν καταλάβατε αυτό. Δεν είμαι καθόλου έτσι, κύριε Κιζουλιέκ. Ευχαριστούμε υποψήφια επίτροπε. Ευχαριστούμε πολύ, υποψήφια Επιτροπέ. Κύριε Κιζιλγιούρεκ, έχετε δεύτερη ερώτηση, συμπληρωματική. Θα συνεχίσω στα ελληνικά, ίσως εννοηθούμε καλύτερα. Πολιτισμικός ρατσισμός είναι μια φράση που υπάρχει σε όλες τις γλώσσες. Στα ελληνικά ονομάζεται πολιτικό ρατσισμός. Στα γερμανικά ρατσισμό. Στα αγγλικά cultural racism. Και μάλιστα έχει τεράστια σημασία γιατί είναι αυτό ακριβώς που ανατρέπει την ετε, ετερότητα στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη μέσα από την ετερότητα όπως συμφωνάμε και οι δύο μας. Όμως πολλές φορές ακούσαμε ότι απέτυχε πολυπολιτισμικότητα στην Ευρώπη. Το έχουμε ακούσει και από την κυρία Μέρκελ από τη Γερμανία και από άλλου ότι απέτυχε η πολυπολιτισμικότητα. Άρα έχει μεγάλη σημασία να υπερασπίσουμε την πολυπολιτισμικότητα. Ερώτημα μου σε εσά είναι τι θα κάνετε για να ενδυναμώσουμε μια λειτουργική πολυπολιτισμικότητα. Ε, Κύριε Σχοινά, απάντησε για ένα λεπτό για την πολυπολιτισμικότητα από το γεγονός ότι ένας Κύπριος Ευρωβουλευτής τουρκοκυπριακής καταγωγής με έναν Ελλαδίτη υποψήφιο αντιπρόεδρο μιλάνε στα ελληνικά στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάτε ψάξτε αλλού. Εδώ δεν θα βρείτε πολιτικό ρατσισμό, ούτε πολιτιστικό ρατσισμό. Εδώ είναι η Ευρώπη, κύριε Ριντουρέκ. Θα κάνουμε τα πράγματα αλλιώς. Thank you very... Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Χόμς Χινέλ. Ε, το πρόφερα σωστά. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σχινά. Ω εκπρόσωπο τη Επιτροπή Απασχόληση Να σα ρωτήσω για τους νέου. Οι νέοι είμαστε η γενιά που έχει την καλύτερη κατάρτιση. Ωστόσο έχουμε πολλή ανεργία, απαράδεκτα υψηλή στην Ένωση. Επίση, η επισφάλεια και τα συμβόλαια περιορισμένου χρόνου αυξάνονται εκθετικά και αφορούν 43% των εργαζόμενων. Μεταξύ αυτών, πολλοί δεν μπορεί να βρει σταθερή εργασία τα συμβόλαια μηδενικών ορών, τα συμβόλαια μερικής εργασίας και τα συμβόλαια που δεν υπόκεινται στην ε, νομοθεσία του εργατικού δικαίου είναι όλο και πιο διαδεδομένα. Πολλές φορές δέχονται ε, συνθήκες ιδιαίτερα επισφαλεί. Κύριε Σχοινά, πώς θα βελτιώσετε την κατάσταση των νέων εργαζομένων, ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση σε μια εργασία αξιοπρεπή, με τις σωστές δεξιότητες και ποιότητας και πώς θα διευρύνετε την κοινωνική τους προστασία. Συμφωνείτε ότι δεν φταίει μόνο η πληροφορική για αυτά τα προβλήματα. Άρα η κατάρτιση δεν είναι η μόνη λύση. Δεν βλέπετε ότι όλα αυτά οφείλονται στο ότι άτομα με τρομερά προσόντα δουλεύουν σε θέσεις πολύ χαμηλής ειδίκευσης και αμοιβή. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Κύριε Χόμς, όντως πιστεύω, πολύ σωστά θέτετε το θέμα, και πραγματικά ε, εντοπίζεται ένα ευρωπαϊκό παράδοξο. Μια αντίφαση. Ποτέ δηλαδή στο παρελθόν, στην ιστορία της απασχόλησης, έχουμε τόσους Ευρωπαίους ε, με θέσεις απασχόλησης. Έχουμε ιστορικό υψηλό απασχόληση. Αλλά το παράδοξο είναι ότι ναι, μεν έχουμε υψηλά ποσοστά, όλο και περισσότερο υψηλά ποσοστά απασχόλησης, έχουμε επίσης πολλές ανισότητες και δυσκολίες στην πρόσβαση και προβλήματα ακριβώς επισφάλειας. Αυτά είναι ουσιώδη προβλήματα και είναι προβλήματα ευρωπαϊκά. Αλλά θα ήταν λάθος πιστεύω εμείς εδώ από τις Βρυξέλλες να πούμε υπάρχει μία λύση κοινή για την κατάσταση των ε, αγορών εργασίας όλων των κρατών μελών. Αυτό που θα κάνουμε με αυτήν την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτό που κάνουμε λοιπόν κάθε χρόνο και σε κάθε χώρα, με πολύ ακρίβεια, είναι το εξή. Λέμε στα κράτη-μέλη, όπου βλέπουμε, είναι σημαντικό να το διευκρινίσω και αυτό, ε, τους λέμε λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, 60% από τις συστάσεις αναχώρα έχουν να κάνουν με τις ε, με την απασχόληση, τις δεξιότητες και την υγεία. Θέματα αρμοδιότητάς μου. Ξέρω λοιπόν ότι η εργασία του εξαμήνου πρέπει να συνεχιστεί και να τη στηρίζουμε παράλληλα. Πρέπει να συνεργαστούμε με τα μέσα που έχουμε, το κοινωνικό ταμείο δηλαδή, ακριβώς για θέματα συμπερίληψης όλων, γιατί εκεί 20 με 25% ακριβώς ε, είναι πόροι για την ε, συμπερίληψη. Και ένα άλλο τμήμα είναι το τμήμα Γκάμπριελ, Ερασμοσύν και επαγγελματική κατάρτιση. Και μέσω αυτών των δυνατοτήτων μπορούμε να προσανατολίσουμε το Ερασμοσύν. Θα πρέπει να μην γίνεται μόνο σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο μαθητεία. Ευχαριστώ για τη συμπληρωματική ερώτηση. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ναι, αλλά τι συνθήκε εργασία έχουν οι μαθητευόμενοι, αυτοί που κάνουν στάζ, τι αμοιβή παίρνουν και τι μαθαίνουν τι εμπειρία έχουν. Γιατί εξακολουθεί να είναι ένα από τα στοιχεία που μας ανησυχεί. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Γιατί οι πρωτοβουλίε που έχουμε, όπω ε, το πλαίσιο ποιότητα για του μαθητευόμενου, δεν έχουν βελτιώσει την κατάσταση. Συμφωνείτε ότι πρέπει να αμείβονται με γραπτό συμβόλαιο. Και τελειώνοντα, ένα άλλο θέμα να αναφερθώ στο όνομα του χαρτοφυλακίου σας. Πολλοί σας είπαν να αλλάξετε το όνομα. Εγώ θα σας έκανα μια πρόταση. Να είναι ο τίτλος σας κάτι που θα πρέπει να είναι η Ευρώπη. Μια Ευρώπη σίγουρη, με αλληλεγγύη και με περισσότερη πρόσδεση ε, στην ε, πολυμορφία και την πολυπολιτισμικότητα της Ευρώπης. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, για το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι συμφωνώ με το περιεχόμενο που προτείνετε. και νομίζω ότι οι δύο ώρες και πάνω που πέρασα εγώ τις πέρασα εξηγώντα ε, πώς εγώ βλέπω την εργασία μου που είναι πολύ παρόμοια με την περιγραφή τη δική σας. Για το θέμα τώρα των μαθητευομένων. Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι υπάρχει περισσότερη συνειδητοποίηση ότι οι μαθητευόμενοι δεν πρέπει να υπόκεινται σε τέτοιες ε, μορφές εργασίας επισφαλής. Αυτό στην ουσία διαστρέφει την έννοια της κατάρτισης. Η μαθητεία έχει έννοια μόνο αν είναι περιορισμένη με πολύ σαφώς ε, καθορισμένης καθορισμένο το επίπεδο των δεξιοτήτων που θα πρέπει να παρασχεθούν και για μένα κάτι που είναι πολύ σημαντικό, αμοιβόμενε. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, για μένα η μαθητεία δεν είναι μαθητεία, είναι κάτι άλλο. Η Επιτροπή νομίζω ότι βελτιώνει κάπως τα πράγματα. Θα συνεχίσω όμως να εργάζομαι με τον Επίτροπο Σμιτ για να γίνει μια αρχή ε, γενικά αποδεκτή. Αυτή η αντιμετώπιση της μαθητείας. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια, κυρία Ρίμπα Ιχινέρ, την Επιτροπή Πολιτισμού και τους Πράσινους. Γεια σας κύριε Σχοινά. Η ελευθερία πολιτιστική, ε, έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια. Ε, φυλακισμοί καλλιτεχνών που έχουν ασκήσει το δικαίωμα έκφρασης τους ε, είναι πολλοί. Και κυρίως ε, η αυτούργη αυτών είναι οι κυβερνήσεις. Ο πολιτισμός είναι σημαντικό εργαλείο διαπολιτικού διαλόγου για να οικοδομήσουμε κοινωνίες που δεν ε, αποκλείουν, που δεν είναι ρατσιστικές, ε, που αγκαλιάζουν όλες τις ιδεολογίες, ε, δεν είναι δυνατόν να λογοκρίνουμε και να καταπιέζουμε την πολιτιστική έκφραση ιδιαιτέρως των γυναικών, των πολιτιστικών μειονοτήτων, των κοινοτήτων ΛΟΑΤ ή των ομάδων που επικρίνουν το σύστημα των αντισυστημικών ομάδων. Έχουμε όλο και μεγαλύτερο, μεγαλύτερο αριθμό δικών εναντίον καλλιτεχνών και λογοκρισιών, ε, ε, επεισοδίων λογοκρισίας. Τι μέτρα θα πάρετε για να ενισχύσετε την πολιτική έκφραση ως μέσο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων. Θα αξιολογήσετε την νομοθεσία των κρατών μέλων που πολλές φορές παραβαίνουν την ευρωπαϊκή, τους ευρωπαϊκούς κανόνες ελευθεριών. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά ο λόγος του κύριου Σχοινά. Κυρία Ρίβα Χινέρ, όλα τα κράτη-μέλη μας είναι δημοκρατίες και έχουν υπογράψει την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ε, συμφωνούν με τις ελευθερίες που περιγράφονται εκεί και ως άτομο αλλά και ως ε, υποψήφιος ε, επίτροπος δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι η πολιτιστική έκφραση ή ε, καλλιτεχνική έκφραση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ρυθμίσεων. Επουδενή δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Η καλλιτεχνική έκφραση και οι καλλιτεχνικές ελευθερίες, η δημιουργική μας δύναμη ε, και ό,τι παράγουν αυτά αποτελούν επίσης τμήμα του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Γι' αυτό είμαστε μοναδικοί και μας ταυμάζουν και ορισμένοι μάλιστα μας ζηλεύουν κιόλας. Νομίζω ότι έχετε στο μυαλό σας κάποια παραδείγματα προφανώς που ίσως να αγνώ. αλλά με δυσκολία θα μπορούσα να φανταστώ ένα δικαστή ε, που θα καταδίκαζε κάποιον για την καλλιτεχνική του έκφραση. Γιατί αυτό το ζήτημα συνδέεται στενά με την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Ε, ούτε εγώ, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να παρέμβουμε ενώπιον των δικαστικών αρχών για να τους υποδείξουμε τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Υπάρχει ο διαχωρισμός των εξουσιών, συνταγματικός διαχωρισμός σε κάθε κράτος μέλος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είμαι διατεθειμένος μαζί με τη Μαρία Γκαμπριέλ και με τις υπηρεσίες μας να εξετάσουμε οποιαδήποτε περίπτωση ε, ή καταγγελία που σχετίζεται με τις ευρωπαϊκές πάντοτε αρμοδιότητες. Θα με ενδιαφέρον να ξέρω τι πραγματικά συμβαίνει και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Mrs. do you have follow-up question? Κύριε Ρίβα Ιχινέρ, συμπληρωματική ερώτηση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Σύμφωνα με πολλέ μη κοινωνικέ οργανώσει, έχει αυξηθεί η χρήση εκ μέρου κυβερνήσεων μέτρων που έχουν ως στόχο να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται για να τιμωρούνται τέτοιου είδους ομάδες όπως αυτές που σας ανέφερα. Στην Ισπανία υπάρχει ο Φαλτόνι, στην Ισπανία ένας ε, τραγουδιστής, ο οποίος ε, για τα λόγια των τραγουδιών του, για τους στίχους, ε, βρέθηκε στη φυλακή, τώρα είναι εξόριστος στο Βέλγιο. Η ίδια η, η, ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κρίνει παράνομο το, ε, το ένταλμα σύλληψής του. Ε, αυτό, αυτού του είδους υποθέσεις επηρεάζουν τις ε, ευρωπαϊκές ε, προδιαγραφές ελευθεριών. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις φυλακίσεων ανθρώπων που απλώς εκφράζονται καλλιτεχνικά. Ο κύριος Σχοινάς, θα επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή. Για μένα η ελευθερία έκφρασης και η καλλιτεχνική δημιουργία είναι καθολική αρχή που μας χαρακτηρίζει. Δεν γνωρίζω την περίπτωση την οποία, στην οποία αναφερθήκατε, αλλά από ό,τι κατάλαβα αυτό έχει σχέση με μια δικαστική απόφαση. Δεν γνωρίζω τις συνθήκες στις οποίες ελήφθη αυτή η απόφαση. Εγώ πάντοτε στην επαγγελματική μου ζωή, ως υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, έχω προσπαθήσει να σέβομαι τον διαχωρισμό των εξουσιών. Αυτό από την εποχή του Μοντεσκιέ ε, είναι μια πραγματικότητα και είναι άλλο ένα από αυτά τα στοιχεία που μας ορίζει, μας καθορίζει και το έχουμε μοιραστεί με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δεν γνωρίζω τις παραμέτρους μια συγκεκριμένης περίπτωση ενός συγκεκριμένου επεισοδίου που προφανώς έχει σχέση με μια συγκεκριμένη δικαστική ερμηνεία και απόφαση. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, κυρία Μπάντινγκ, από την Επιτροπή Πολιτισμού, από την ομάδα Ρινιού. Κύριε Σχοινά, σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας. Είναι μεγάλη μου χαρά να ακούω να επαναλαμβάνετε με τέτοια πειθό ότι θα προστατεύσετε την ποικιλομορφία στην Ευρώπη. Είμαι φιλελεύθερη. Το λέω ευθύ εξ αρχή. Και δεν θέλω καθόλου να υπάρξει επιθετική πολιτική για τι ταυτότητε του κόσμου. Όμω, όπω και άλλοι εδώ, μου αρέσει Ιταλικό πολιτισμό, Ελληνικό, Γερμανικό πολιτισμό, ακόμη και Βρετανικό. Ναι, μέχρι και αυτό. Δεν θέλω κανεί εκτό ε, τη Ευρωγιάλα όμω να πιστέψει ότι κανεί από εμά επιμένει ότι υπάρχει μόνο ένα ευρωπαϊκό τρόπο ζωή και για την πρώτη μου ερώτηση. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω για τι πρακτικέ διαθετήσει τη θέση σα. Είστε υπεύθυνο για την επαγγελματική και τη διαβίου μάθηση και την διασυνοριακή μάθηση. Αναφέρατε το Erasmus Συν πολλέ φορέ. Πώ σκοπεύετε να συνεργαστείτε με άλλου επιτρόπου, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι η ευρωπαϊκή επίδραση στο εκπαιδευτικό σύστημα θα προάγει την ευρωπαϊκή πολιτιστική ποικιλομορφία καθώ και την κρίσιμη, αλλά λιγότερο αντιφατική ε, ψηφιακή καινοτομία καθώ και τι επαγγελματικέ αρμοδιότητε που, χρε... Ε, ε, που χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Μπούντινγκ ε, για το πρώτο μέρος της ερώτησής σας. Καταλαβαίνετε προφανώς ότι συμφωνούμε. Για το δεύτερο σκέλος. Για τα όρια των αρμοδιοτήτων μου και πώς θα λάβω θέση εγώ ίδιος. Να σας πω κάτι που έχω ζήσει. Όταν ετοιμαζόμουν για την ανταλλαγή αυτή απόψεων και με ενημέρωναν οι υπάλληλοι της Επιτροπής. Τη στιγμή που θα με ενημέρωναν για τις δεξιότητες, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τα ψηφιακά, ήμασταν 55 άνθρωποι γύρω από το τραπέζι ξαφνικά. Και είπα, τι έγινε και γίναμε τόσοι πολλοί. Και κάποιος έδωσε μια ωραία απάντηση διότι ιστορικός και παραδοσιακός αυτό ε, γινόταν εκεί και ο τάδε τμηματάρχης πήγε την υπηρεσία από εκεί εκεί και στην τάδε και γενική διεύθυνση. Ε, αυτό είναι ένα παράδειγμα για να σας εξηγήσω. Γιατί η κυρία Φοντερ Λάιεν θεώρησε ότι χρειάζεται αντιπρόεδρο που πολιτικό θα λογοδοτούσε σε εσά και θα ήταν υπεύθυνο ε, έναντι εκείνη για να συνδυάσει προστιθέμενη αξία από αυτήν την πληθώρα οργανισμών, υπηρεσιών, φορέων. Εγώ χαίρομαι πολύ για αυτή τη δουλειά. Πραγματικά μου προκαλεί ενθουσιασμό, διότι δεν μ' αρέσει ο καταγερματισμός δεν θέλω να πρέπει 50 άτομα να με ενημερώνουν για ένα χαρτοφυλάκιο και χαίρομαι που πολλά τα θέματα που συζητήσαμε, η διαβίου μάθηση, η ενέργεια των νέων, οι επαγγελματικέ δεξιότητε, η βελτίωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι παντού σκορπισμένα στην Επιτροπή. Δεν το θέλω αυτό. Ο ρόλος μου λοιπόν, μαζί με τον Επίτροπο για τις θέσεις εργασίας, μαζί με τον Επίτροπο για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ε, παιδεία, μαζί με τον Επίτροπο για την ισότητα, μαζί με τον Επίτροπο για την υγεία Όλα αυτά μπορούμε να τα συναρμόσουμε. Και γι' αυτό έρχομαι και, σας, και θα έρχομαι να σας εξηγώ πώς τα πήγα. Πέτυχα, απέτυχα, αλλά θα έχετε εμένα και όχι 50 επιτρόπους. Ευχαριστούμε. Έχετε επιπλέον ερώτηση κύριε Μπάντινγκ. έχει να κάνει και πάλι με τον τίτλο του χαρτοφυλακίου σας. Λυπούμε. Αλλά ε, σίγουρα το ξέρατε και το συζητήσατε με την der Leyen ε, πριν έρθετε εδώ. Το περιμένατε αυτό που αντιμετωπίζετε. Όμως πραγματικά βλέπετε όλη αυτή η αίθουσα από την δεξιά και την αριστερά, από τη Λίμπε και την Κουλ ε, τις δικοινοβουλευτικές επιτροπές, από όλους να δέχεστε αμφιβολίες. Εγώ δέχομαι ότι αυτά που λέτε είναι καθαρά και ξάστερα και είμαι στο πλευρό σας. Όμως το ο τίτλο του χαρτοφυλακίου είναι κακό. Πραγματικά μην είστε υπεροπτικό, ούτε να τηρείτε αμυντική στάση. Πηγαίνετε στην Ursula von der Leyen και ζητήστε να επαναδιατυπώσετε τον τίτλο σα. Εγώ θα έλεγα κάτι σαν Α προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Κάτι τέτοιο. Κάτι που να μην. Εάν εμεί ανησυχούμε, τι θα πούν οι πολίτε. Θα ανησυχήσουν περισσότερο τη δική τους προσοχή θα τραβήξει όλο αυτό. Μην είστε ε, αλαζόν και πραγματικά ε, υποσχεθείτε ότι θα περάσετε τουλάχιστον ένα μισάωρο να το συζητάτε με την Ursula von der Leyen. Ευχαριστούμε κυρία Μπάντινγκ. Για ένα λεπτό κύριε Σχοινά θέλετε να το απαντήσετε. Να σας πω ότι είναι τιμή μου. Τιμή μου που σας έχω στο πλευρό μου. Αυτό είναι ήδη από μόνο το επιτυχία. Δεύτερον, το είπα και στη Σόφη Ιντβελτ. Για το που βρισκόμαστε Πραγματικά το λέω. Δεν θεωρώ ότι υπήρξε άλλα ζώνα. ήμουν, ζητώ συγγνώμη. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το δούμε στα πλαίσιο, το συνολική εικόνα του τι είπε, εξήγησε η υποψήφια πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ψηφίσατε και πιστεύω ότι καθησύχασε τις ε, αμφιβολίες σας, τις διασκέδασε. Σέβομαι πλήρως όλα τα επιχειρήματα που διαμορφώνουν τη σημερινή μας συζήτηση. Τα σέβομαι πλήρως. Και είχα την ευκαιρία να πω ότι σε αυτή την ιστορία έρχομαι με μια θετική στάση και θετική οπτική γωνία. Δεν θέλω να το χρησιμοποιήσουν αυτό και να το εκμεταλλευτούν οι εξτρεμιστέ. Θέλω να μείνουμε στη θετική πλευρά των πραγμάτων. Λέτε να πάω πίσω στην πρόεδρο τη Επιτροπή και να τη το πω. Μα σα είπε ήδη ότι στην Ευρώπη συζητάμε και εν τέλει συμφωνούμε. Αυτό σας είπε. Αυτό το έγραψε και στην επιστολή της. Αυτά. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση μου. Ισαβέλ Μπενχουμέα Μπενχουμέα, Επιτροπή Πολιτισμού, ε, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σχοινά. Τελευταία ερώτηση. Καθ' όλη τη συζήτηση συζητήσαμε για τη το φιλόδοξο θεματολόγιο που έχετε θέσει για την εκπαίδευση, όπου λέτε καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, να αντιμετωπιστεί το θέμα των μαθητών που καταλήγουν το σχολείο, διαβίου κατάρτιση, τα άτομα άνω των 50 που έχουν ε, προβλήματα πρόσβαση στην αγορά εργασία και μιλήσαμε και για την επαγγελματική κατάρτιση, σημαντική πρόκληση. Αλλά για να προστατεύσουμε τον ε, τρόπο ζωής μας και τις ευρωπαϊκές αξίες είναι σαφέ ότι αυτό που υπερασπιζόμεθα είναι η ελευθερία, το κράτο δικαίου και πάνω απ' όλα ότι η Ευρώπη να δίνει ευκαιρίε σε όλου. Και τι ευκαιρίε τι δημιουργούν οι επιχειρηματίε, αυτοί που επενδύουν, που δημιουργούν επιχειρήσει. Θα ήθελα να μου πείτε, όταν μιλάτε για εκπαίδευση, πώ θα δημιουργήσουμε επιχειρηματικό πνεύμα. Τι πρέπει να κάνουμε στην Ευρώπη για να υπάρχουν περισσότεροι επιχειρηματίε που να δημιουργούν ε, ε θέσεις και ευκαιρίε για όλου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέχουμε. Όντως. Θέτεται το εξή θέμα. Λέμε ότι όλη μας η εργασία για την κατάρτιση των πολιτισμό, εκπαίδευση, για την νεότητα, δεν κάνουμε μία ενιαία αγορά εκπαίδευσης και δεν χρειάζεται να κάνουμε γιατί τα κράτη-μέλη έχουν ε, αρμοδιότητες για τα θέματα αυτά. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Θέλουμε να συμβάλλουμε. Θέλουμε να καταρτήσουμε τους νέους μας, τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες μας. Για να κάνουν τα δύο που αναφέραμε προηγουμένως. Πρώτα απ' όλα να έχουν καλύτερες δεξιότητες, να φτιάξουμε τη γέφυρα ανάμεσα σε αυτό που, όπου έχουμε λήψεις και τους ε, εργαζόμενους και τη βελτίωση των δεξιοτήτων. Να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας που έχουν μείνει στο περιθώριο της τεχνολογικής προόδου για να προχωρήσουν. Συμφωνώ. Εάν βοηθήσουμε έτσι τους εργαζόμενους μας, βοηθάμε και την οικονομία μας και την κοινωνία μας. Δεν το κάνουμε για μας ή για αυτούς. Έχει απευθεία σχέση, δημιουργεί απασχόληση, δημιουργεί ανάπτυξη, πλούτο αυτό το επιχειρηματικό πνεύμα. Να κάνουμε δηλαδή την κατάλληλη κατάρτιση για να έχουμε επιχειρηματίες δεν είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε απευθεία. Δεν μπορούμε να του πούμε έτσι θα γίνει επιχειρηματία. Πρέπει να του δώσουμε την κατάρτιση, τα πτυχία, τι γλωσσικέ γνώσει για να μπορέσουν να δημιουργήσουν θέσει εργασία. Και πολλά προγράμματά μα, όπω το πρόγραμμα επενδύσεων Juncker, όλα τα προγράμματα επενδύσεων μέσω του Horizon 2020 στην τεχνολογία ακριβώς θα βοηθήσουν να δημιουργηθούν επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία συμπληρωματική ερώτηση, κυρία Μπενχουμέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Εγώ βασίζομαι στο ότι ορισμένοι γεννιούνται επιχειρηματίες, αλλά άλλοι γίνονται. Για να γίνουν επιχειρηματίες, δεν θα επιβάλλουμε σε κανένα να γίνουν επιχειρηματίες. Όχι. Αλλά πρέπει να έχουμε τη φιλοδοξία να υπάρχουν όλο και περισσότεροι επιχειρηματίε. Περισσότερα άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν ευκαιρίε, πλούτο, θέσει εργασία. Γιατί αυτοί θα πληρώσουν τους, τους φόρους για να διατηρηθεί το κράτος ευημερίας που είναι και αυτό χαρακτηριστικό της Ένωσης. Γι' αυτό επιμένω στην ερώτησή μου. Γιατί δεν είναι στην επιστολή καθηκόντων. Εάν υπάρχει η βούληση όταν μιλάμε για εκπαίδευση, να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να εργαστούμε για να δημιουργήσουμε ενθουσιασμό στους νέους, τη φιλοδοξία. Να πούν, μπαμπά, μαμά, θέλω όταν μεγαλώσω να γίνω επιχειρηματίας. Όχι, δεν, δεν είναι στην επιστολή που μου έστειλε η κυρία Φόντε Λάιν και δεν είναι, δεν αναφέρεται συγκεκριμένα ο στόχος που να αναφέρεται ρητά στις δυνατότητές μας. Αλλά έχουμε ένα ολόκληρο φάσμα δυνατοτήτων που μας επιτρέπει. Πρώτον, να εντοπίσουμε ποιες δεξιότητες μας λείπουν. Αυτό από μόνο του βοηθάει τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις κλήσεις τους. Αν ένας νέος, ένας φοιτητής πραγματικά θέλει να γίνει επιχειρηματία, τότε πρέπει να μπορούμε να του πούμε, κοίταξε, αυτή είναι μία οδός για να το επιτύχεις. Αλλά δεν μπορούμε σε κανένα να επιβάλλουμε να μάθει να γίνει επιχειρηματίας. Αυτό πρέπει να είναι ένα πιο πολύ ευρύ καθήκον, όπου πρέπει να συνεργαστούμε και εμείς μεταξύ μας ως Επίτροποι και εσείς ε, και τα κράτη-μέλη φυσικά. Ευχαριστώ πολύ κλείνουμε και το δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ που με ακούσατε και θα δώσω την προεδρία στον κύριο Λοπεθαγγιλάρ. Ολοκληρώσαμε 25 ερωταποκρίσει των 5 λεπτών, παρόλο που ξεπεράσαμε για λίγο το χρόνο μας και πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της κοινή συνεδρίασης. Πριν όμως, πριν κλείσουμε, έχετε τη δυνατότητα να πείτε κάποια τελευταία λόγια, πέντε λεπτά, ο λόγος στον κύριο Σχοινά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι αργά ήδη. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ πλούσια και πλατιά συζήτηση, σφαιρική, που κατέδειξε ένα πράγμα. Χωρίς καμία αμφιβολία, η προσήλωση όλων σας είναι πάρα πολύ υψηλή. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πριν ζητήσω την εμπιστοσύνη σας, ε, θέλω να λάβετε υπόψη πως το έργο που μου εμπιστεύονται είναι κάτι καινούριο. Είναι μια καινούρια θέση εργασία. Ε, που έχει τη δική της περιγραφή. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί χρειάζεται αυτή, αυτό το καινούριο πόστο στην καινούρια κομισιόν. Και η απάντηση πιστεύω ότι είναι και ελπίζω να σας έπεισα ότι παρόλο που το πόστο είναι καινούριο, τα προβλήματα είναι παλιά. Και είναι πολύ ριζωμένα στο πώς έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν η κοινωνία μας. Έχει οργανωθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με μια συγκεκριμένη λογική, με επιμερισμούς και κατακαιρματισμούς και με τη βοήθεια των επιτρόπων που θα συνεργαστούν μαζί μου και τους, θα τους συντονίσω, θα τους καθοδηγήσω, στόχος είναι όχι μόνο να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση των όσων σας υποσχεθήκαμε τον Ιούλιο, αλλά, πολύ πιο σημαντικό, όλες αυτές τις πτυχές να τις ενοποιήσουμε σε ένα ενιαίο αφήγημα καλών πρακτικών, ε, ποικιλομορφίας, πλούτου, αρχών, ικανοτήτων, έτσι ώστε να οικοδομήσουμε πραγματικά ε, μια ανθεκτική και ανεκτική Ευρώπη για το μέλλον. Ελπίζω ότι καταλαβαίνετε ποια θα είναι η δική μου μικρή συνεισφορά. Γι' αυτό θα πολεμήσω και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να το πετύχουμε μαζί τα επόμενα πέντε χρόνια. Ευχαριστώ. Εμεί Να σας ευχαριστήσουμε κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε, κύριε Σκινά, και να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη για την υψηλή προσέλευσή τους σε τέτοια προχω... προκεχωρημένη ώρα μέσα στη μέρα για να ολοκληρώσουμε αυτήν την ε, μακροσκελέστατη συνεδρίαση πάνω από τρεις ώρες, να πούμε ότι έχετε αναλάβει ένα χαρτοφυλάκιο πραγματικά ε, γεμάτο από υποσημειώσεις, ερωτηματικά και για να μην πω και ενστάσεις. Γιατί υπάρχει ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, αλλά το να δουλεύει κανείς τόσο αργά καθόλου δεν συνάδει με τους κανόνες για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Και το δεύτερο που θα έλεγα είναι ότι ναι, Μπορεί να υπάρχει ευρωπαϊκό τρόπο ζωή, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα και μόνο. Ούτε μια εκδοχή που πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλου. Ο ευρωπαϊκό τρόπο ζωή βασίζεται στο να είναι ανοιχτό, να επιτρέπει τη συμμετοχή όλων, να μπορεί να δεχτεί την ποικιλομορφία και τον πλουραλισμό, την πολυφωνία. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους που παρακολούθησαν αυτή τη συζήτηση και να, ανακοινώσω ότι εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και η συμπρόεδρος θα συγκαλέσουμε την συνεδρία των συντονιστών για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ως δι την έκβαση της ακρόασης, της συζήτηση που μόλις είχαμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε κύριε Σχοινά. Καλή τύχη. Oh, και εγώ θέλω να πω δύο κουβέντε. Ε, πρώτα απ' όλα ευχαριστήσει προ τον κύριο Σχοινά. Ε, Όπω περιμέναμε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και θερμή συζήτηση και πρέπει να πω ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις και επίσης και στους συναδέλφους ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις που θέσατε διότι και εσεί ήσασταν ε, αναπόσπαστο μέρο της απόψινής συζήτηση. Ευχαριστώ και τον συμπροεδρό μου, τον Χουάν ε, Λόπε Αγγιλάρ, για την άριστη συνεργασία μα στην ακρόαση αυτή. Ευχαριστούμε και τι γραμματείες, του συνεργάτε μα για τη διοργάνωση, γιατί όλα πήγαν όπω έπρεπε και πολύ καλά. Όπω ξέρετε, επόμενο καθήκον μας είναι να αξιολογήσουμε, να αποτιμήσουμε όσα ακούσαμε απόψε το βράδυ. Και θα σας ζητήσω να είστε από τις 10 ε, παρατέταρτο μαζί με τους και, και, 10 και 4 να είστε με τους συντονιστές της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ στο 1G3 στο κτίριο ASP Αλτιέρο Σπινέλη. Παρακαλώ όλοι, όλοι οι συντονιστές να με ακούσετε και οι υπόλοιποι κάπως ησυχάστε για να παρακολουθείτε τι λέω. Ένα λεπτάκι την προσοχή σας παρακαλούμε. Δεν ολοκληρώσαμε ακόμα. Παρακαλώ συνάντηση των συντονιστών στις 10 και 4 στο ASP 1G3. Παρακαλώ όλοι οι συντονιστές της ΛΥΜΠΕ και της ΚΑΛΤ να, Κουλτ να είστε εκεί για να ολοκληρώσουμε εγκαίρως τη δουλειά μας απόψε. Η Επιτροπή Απασχόλησης και ο συμμετέχουσα υποσκεκλημένη Επιτροπή θα εκπροσωπείται με ένα από τους Προέδρους της. 10 και 4 στο ASP 1G3. 3G G3. Hello. I just forgot to say thank you also to the... Ξέχασα να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς μας για τη δουλειά τους απόψε. Δεν είναι εύκολη η δουλειά τους και μια, ένα μικρό χειροκρότημα για τις κυρίες και τους κυρίους της καμπίνες που το επέτρεψαν αυτό σε όλες τις γλώσσες. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.